Colleagues, με το επόμενο σημείο της μέσης διάταξης. Δεύτερη εξέταση του σχεδίου ψηφίσματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. 406 τροπολογίες. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ενίσχυση της εταιρικής ε, σχέσης, η θέση της Ευρωπαϊκής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις πρόοδου. Ε, ο συνεισηγητής, ο κύριος Σάριους Βόλσκι, ε, θα μας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινωνία και ο κύριος Παντζέρη επίσης. Ε, θέλω να καλωσορίσω τον Φίλιπ Δημητρόφ που είναι ο πρέσβης ε, που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της Γεωργία, πρέσβης στην Τυφλίδα. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάριους Βόλσκι, συνεισηγητή για την Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία. Ευχαριστώ. Πρόσφατα κάναμε την πρώτη ανάγνωση της εκθεσής μου. Ε, δεν έχει περάσει πολύ καιρός. Ε, 460 τροπολογίες έχουμε. Ευχαριστώ όλους όσους τη συνέταξαν. Εγώ και ο κ. Παντσέρη προσπαθήσαμε να τις διαβάσουμε καταρχάς και προσπαθήσαμε συνεχεία να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Δεύτερη παρατήρηση. Στην ε, πολιτική ε, γειτονίας προς Ανατολάς τα πράγματα κινούνται. Ε, έχουμε πολλές αλλαγές. Ακούσαμε και τα, την πρωινή συζήτηση στα πλαίσια της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας με την Ουκρανία. Λόγω των γεγονότων, ίσως υπάρχουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε όλα τα στοιχεία επιτάπητος, μπορεί το χρονοδιάγραμμα να επιβραδυνθεί. Αλλά ο πρόεδρος Μπροκ θα αποφασίσει τελικά γι' αυτό. Θα δούμε τι θα, εξέλιξεις θα έχουμε. Το βασικό θέμα είναι πότε η Ουκρανία θα συμμορφωθεί με όλες τις προϋποθέσεις. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Και εμείς θα πούμε συνεχεία στην έκθεσή μας το κατά πόσον συνιστούμε ή όχι την ε, υπογραφή της συμφωνίας. Επομένως η πολιτική γειτονία προς Ανατολάς δημιουργεί κάποια προβλήματα. Και κύριε Παντζέρη, καταλαβαίνετε ότι η στάση αυτή τη πλευρά, τη Ουκρανίας δηλαδή, θα επηρεάσει και τη θέση μα στη συμφωνία. Είχαμε τρει ε, διαφορετικέ συναντήσει των σκιωδών εισηγητών. Μία για το γενικό τμήμα τη έκθεση και δύο χωριστέ συνεδριάσει των σκιωδών. Ε, μία για την ανατολική πλευρά, του ανατολικού γείτονε και μία για του νότιου. Ευχαριστώ τον κύριο Παντσέρη για την θαυμάσια συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμή, για την ε, κοινή έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία προ Ανατολά και προ Νότο. Οι τροπολογίε είναι πολύτιμε ω προ την ουσία του, αλλά συχνά επαναλαμβάνουν οι μεν αυτά που λένε οι δε. Ορισμένε είναι, είναι και εκτό θέματο. Όλα αυτά λοιπόν τα λαμβάνουμε υπόψη μα και όσε είναι εκτό θέματο θα τι απορρίψουμε, χωρί να αξιολογήσουμε το περιεχόμενό τους. Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού με τον κύριο Παντζέρη ότι θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες που εμπλουτίζουν την έκθεση με νέα στοιχεία, με ουσιαστικά στοιχεία. Κάποιες δηλαδή, και ελπίζουμε και αυτοί που τις υπέβαλαν, ε, θα δεχτούν και θα καταλάβουν το γεγονός ότι πρέπει να τις απορρίψουμε, τις τροπολογίες τους. Για την ανατολική πολιτική γειτονία, εγώ είμαι γενικά αισιόδοξο για το τελικό αποτέλεσμα. Και αν υλοποιηθεί το αισιόδοξο σενάριο, σε ό,τι αφορά τις ε, προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους, αυτή η έκθεση μπορεί να έρθει την κατάλληλη στιγμή και να λέει αυτά που μπορεί να υλοποιηθούν στη Σύνοδο Κορυφής ε, του Βίλνιους. Τι εννοώ δηλαδή. Και Εκεί καταλήξαμε στις πρωινές μας συζητήσεις με τον κύριο Σάλιβαν, ότι αν τα πράγματα πάνε κατευχήν, όπως ελπίζουμε και θέλουμε, και ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο για την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, με την, μετά την υπογραφή, αυτή η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει μία φράση, μία παράγραφο που θα σέβεται την ε, προϋπόθεση όχι της συνθήκης, αλλά αυτή της ε, συμφωνίας κυρίων που έχουμε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δηλαδή τι εννοώ, η επικύρωση, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Και εμείς μπορούμε να πούμε λοιπόν σε αυτήν την παράγραφο ότι θέλουμε η επικύρωση να γίνει πριν από το τέλος της νομοθετικής θητείας ε, του Κοινοβουλίου. Το αργότερο την Άνοιξη. Αλλά επειδή η Ουκρανία έχει, βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θέλουμε να δώσουμε το πράσινο φως στο Συμβούλιο να εφαρμόσει πλήρως και χωρίς περιττές καθυστερήσεις, κυρίως το εμπορικό κομμάτι της συμφωνίας, προσωρινά, νωρίτερα. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ ξανά τους συντάκτες των τροπολογιών και τον συνεισηγητή μου για τη θαυμάσια συνεργασία. Ευχαριστώ Γιάτσεκ. Και τώρα ο κύριος ε, Παντζέρη που θα μας μιλήσει για την νότια διάσταση της ε, πολιτικής γειτονίας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ βεβαίως τον Σάριος Βόλσκι για το γενικό τμήμα. Τα έχουμε βρει, έχουμε συμφωνήσει. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Πρέπει να συστηματοποιήσουμε και τις διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούμε για να τις χρησιμοποιούμε με, με τον ίδιο τρόπο για το κοινό πάντα τμήμα. Σε ό,τι αφορά την νότια διάσταση της πολιτικής γειτονίας, υπάρχουν μια σειρά τροπολογίες που υποβλήθηκαν και που αναφέρονται σε σημαντικές δηλώσεις της Βαρκελόνης, ε, του Παρισιού, διάφορες ε, συστάσεις και ψηφίσματα και δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα να δεχτούμε αυτές τις τροπολογίες που μιλάνε για αυτές τις δηλώσεις. Όπως και κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται Ε, σε διάφορες αρχές. Και για το ότι οι, πολιτικές, ε, οι ευρωπαϊκές πολιτικές γειτονίας ε, προς όλες πρέπει να είναι ισορροπημένες και προς Ανατολάς και προς Νότο. Ορισμένε τροπολογίε αναφέρονται στην ανάγκη να λάβουμε υπόψη μας τις φιλοδοξίες των λαών του αραβικού κόσμου ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση του κράτους δικαίου, κανένα πρόβλημα. Αυτές οι τροπολογίες βεβαίως μπορούν να γίνουν δεκτές. Βεβαίως πρέπει να τις συστηματοποιήσουμε αυτές τις τροπολογίες. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που μιλάνε πάντα για την νότια διάσταση μόνο. Και εδώ προσπαθούμε απλώ να συστηματοποιήσουμε τις τροπολογίες ώστε να μην ξαναλένε τα ίδια. Τώρα, οι στόχοι τη πολιτική γειτονία που αναφέρονται στο, σε μια αιτιολογική σκέψη από την 73 έως την 84 για τη δημο, δημοσίευση της έκθεσης προόδου και του 2012, συμβαστικές τροπολογίες, θα γίνουν για, την, για άλλες παράγραφοι το, της αιτιολογικής σκέψης, ε, για τη νέα πολιτική γειτονία και παράγραφος 4 για την υποστήριξη της ε, δημοκρατικής μετάβασης και την εμπλοκή της κοινωνία ε, κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των μειονοτήτων κτλ. Όλες αυτές δηλαδή τις έννοιες που έχουν εκφράσει τροπολογίες θα τις λάβουμε υπόψη μας. Και υπάρχει και μια ομάδα τροπολογιών από την, για την παράγραφο 5 έως 13, 144 μέχρι την 2.74 ε, που αφορούν την ανατολική διάσταση και βεβαίως ο συνεισηγητής μου θα μιλήσει για αυτές. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νότια διάσταση τώρα, θα κάνουμε ένα συμβιβασμό για την ε, παράγω που μιλάει για την ε, οργάνωση της Task Force Ο στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να υπογραμμίσει ότι το κοινοβούλιο μας πρέπει να εμπλακεί στην ε, δημιουργία αυτής της Task Force. Και στο ψήφισμά μας για την Ισία του 2011 λέγαμε και ζητούσαμε από την ύπατη εκπρόσωπο να δημιουργήσει αυτή την Task Force. Και επομένως τώρα αυτή η εμπειρία ε, θα πρέπει να ε, επεκταθεί και στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα μια άλλη, ένας Θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση σε αυτές τις χώρες. Θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη. Θα υποστηρίξω λοιπόν αυτές τις τροπολογίες και θα υποστηρίξω και τις τροπολογίες που μιλάνε για την προώθηση μιας πραγματικής περιφερειακής ολοκλήρωσης, πάντα για την νότια διάσταση. Επίσης, υπάρχουν πολλές τροπολογίες, πολύ σύντομα το λέω αυτό, που αφορούν τις επιμέρους χώρες. Επ' αυτών των τροπολογιών Πρέπει να πω ότι επειδή γράψαμε λίγα πράγματα για τις επιμέρους χώρες, προέκυψαν όλες αυτές οι πολλές ε, τροπολογίες. Κάθε φορά έτσι γίνεται. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να πούμε πολλά, εξού και οι πολλές τροπολογίες. Για την Αλγερία, για την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Θα τις λάβουμε υπόψη μας. Φυσικά κάποιες από αυτές δεν μπορώ να τις δεχτώ. Εξάλλου το, τη συζητήσαμε και σήμερα το πρωί με τους ενδιαφερόμενους. Ε, όταν συζητήσαμε την έκθεση Τάνο, ειδικά για το Μαρόκο κτλ. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση πολύ συγκεκριμένη των επιμέρους τροπολογιών στις διάφορες επαφές που θα έχουμε με τους σκιώδες εισηγητές, ούτως ώστε να βρούμε μία συνεπίθεση για αυτές τις συγκεκριμένες ε, τροπολογίες που αφορούν τις επιμέρους χώρες. Νομίζω ότι μπορούμε να δουλέψουμε άνετα και μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Starting with the intervention of the members and of shadow reporters, I would like as I... Θέλω να πω στην αρχή ότι ο κ. Φιλίπ Δημητρόφ, πρόεδρος, ε, συγγνώμη, πρέσβης στην Τυφλίδα, θα μας πει δύο λόγια για τη Γεωργία. Πριν, ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Φυσικά ρίξα μια ματιά στο σχέδιο ψηφίσματος και για την αναφορά στη Γεωργία και τις, τα επιτεύγματα, αξιόλογα επιτεύγματα σε σχέση με τη Γεωργία τα τελευταία δέκα χρόνια. Πράγματι, όποιος είχε πάει στη Γεωργία πριν από αυτά τα χρόνια μπορεί να διαπιστώσει αυτή τη σημαντική διαφορά. Το ερώτημα είναι φυσικά πόσο αμετάκλητα είναι όλα αυτά. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια κοινή τάση που και αναφέρεται σε σχέση με τις τελευταίες ε, σφιγμομετρήσεις, ε, βολιδοσκοπήσεις για έντονη στεναρή υποστήριξη της προσέγγισης προς την Ευρώπη. Έχουμε την αντιπολίτευση που είναι η φιλική προς την Ευρώπη και προς την Δυτική Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις ε, και από πλευρά των αρμοδίων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό παρόλα αυτά να δούμε ποια θα είναι τα βήματα και οι κινήσεις από πλευρά των Ευρωπαίων ώστε να μην διαβρωθεί αυτή η τάση, αυτή η προσέγγιση της Ευρώπης. Λέγοντας αυτό ότι θέλω να πω ότι ανησυχούμε σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή αυτή. Στη Γεωργία όμως δεν ήταν εφικτό να ασκηθεί κάποια πίεση εκ των έξω στην Γεωργία με μεγάλο ποσοστό της επικράτειας που έχει αποσχιστεί από τη χώρα αυτή είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με την επιρροή που μπορεί να ασκηθεί από πλευράς του εξωτερικού προς τη χώρα αυτή δεδομένης αυτής της κατάστασης. Οι κίνδυνοι θα βρίσκονται μάλλον στην εσωτερική πολιτική ζωή και τις ε, δυναμικές τάσεις που θα εξελίσσονται και που πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγης. Για αυτούς τους λόγους δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναμένουμε κάποιες εκπλήξεις πριν από σύνοδο κορυφής του Βίνιους. Και πραγματικά η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι ένας ε, πάρα πολύ έντονα υποστηρίχθηκε πολύ έντονα από πλευράς των προσπαθειών που καταβλήθηκαν και αναφέρθηκε σε σχέση και με το ψήφισμα για γοργή υπογραφή και απελευθέρωση από τις θεωρήσεις διαβατηρίων ιδιαίτερης σημασίας για το ότι θα πρέπει να μπορέσουν να υπάρξουν θετικές προτάσεις ώστε να ενισχυθούν αυτές οι προδιαγραφές. Όπως ανέφερα υπάρχει η πολιτική δυναμική των πραγμάτων. Βρίσκεται υπό συγκεκριμένη συγκυρία η χώρα για τις προεδρικές εκλογές. Θα έχουμε υποψηφίους από το κυβερνών κόμμα, από την φιλοδυτική αντιπολίτευση και από την αντιπολίτευση που ας το πω με πολύ ήπιο τρόπο τρόπο διατυπώνοντας την περιγραφή αυτή είναι εκείνη η οποία δίνει ε, αρνητικά μηνύματα κατά του ΝΑΤΟ και αρνητικές τοποθετήσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το ότι συγκεκριμένοι συμβιβασμοί θα πρέπει να αναζητηθούν, αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τα προβλήματα στην περιοχή αυτή. Όμως ταυτόχρονα είχαμε και τον Πρωθυπουργό που ανέφερε ότι πρόκειται να αποχωρήσει και αναπόφευκτα όλα αυτά τι θα σημαίνουν. Θα σημαίνουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τη δομή και ίσως ε, και διάλυση του κυβερνώντος ε, κόμματος που είναι ένα συνονθήλευμα και πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά του σύνεγγυ στην κατάσταση και να υποπτεύσουμε για τον κίνδυνο ιδιαίτερα εκείνων των φιλοδυτικών στοιχείων σε αυτή τη συμπολίτευση που έχουμε συνηθίσει να τους, βρίσκουν, να τους συναντούμε εδώ στις ε, Βρυξέλλες που ίσως δεν θα μπορέσουν να διατηρηθούν επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην πολιτική σκηνή. Όμως το πιο σημαντικό θέμα παραμένει παραμένει. Παραμένει ότι θα υπάρξει μια σημαντική φιλοδυτική πολιτική τάση στη Γεωργία και για αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο φορέας αυτής της τάσης είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης σε πρώην κυβερνητικό κόμμα θα υπάρξουν φυσικά αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι εν συντομία πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προφανή μηνύματα και στοιχεία που δείχνουν ότι γίνονται προσπάθειες να καταστραφεί αυτή η τάση, αυτό το κόμμα. Είχαμε και μια έκθεση που παρουσιάστηκε κατά τέτοια την Κυριακή υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά είναι ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο που δείχνει ποιες ήταν οι ελλείψεις ε, της παλαιότερης κυβέρνησης αλλά και της νη κυβέρνησης ε, συντάσσοντας ε, συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει και τι δεν επιτρέπεται να είναι αποδεκτό και έγινε από έναν ειδικό υπεύθυνο για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Φιλοδυτικές δυνάμεις στην Γεωργία πρέπει να παραμείνουν εκεί στην θέση τους. Και αυτό με οδηγεί πάλι στη γραμμή έναρξης όπως ξεκίνησα. Η αναφορά στο σχέδιο ψηφίσματος για την αξιοπρόσεκτη πρόοδο που επετέχθη στην Γεωργία σε σχέση με την περίοδο αυτής της δεκαετίας συγκρίνοντας με το τι υπήρχε πριν από αυτά τα δέκα χρόνια οφείλεται σε σχέση με τις προσπάθειες που έγιναν. Είναι σημαντικό ότι γίνεται η προσπάθεια να καταστραφεί τώρα αυτό το κόμμα, να διαλυθεί και αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται ένα κίνδυνο της καταστροφής αυτού του κληροδοτήματος αυτού του κόμματος, μια σημαντική τάση για αυτή τη χώρα, μια σημαντική φιλοδυτική φιλοευρωπαϊκής τάσης που δημιουργήθηκε και ενδυναμώθηκε μετά την περίοδο των ε, ταραχών και όλα αυτά θα πρέπει να τα θυμόμαστε σε σχέση με τη Γεωργία. Φυσικά θα πρέπει να δούμε ότι το πλαίσιο δράσεώς μας ε, έχει και συγκεκριμένους περιορισμούς. Όμως σε σχέση με ένα τέτοιο ψήφισμα όπως αυτό του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να βαίνει προς την ορθή κατεύθυνση με τα όσα εμπεριέχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μητρόφο. Κυρίως ο κύριο θέλει να ρωτήσει κάτι κάποιο σχόλιο παρακαλώ. Ναι, έχω δύο ερωτήσεις προς τον πρέσβη παρακαλώ. Ήδη η κατάσταση στη Γεωργία τον Αύγουστο το 2008 μας ξάφνιασε. Θυμάμαι ότι τον Ιούνιο στην ΑΦΕΤ ψηφίσαμε ένα ψήφισμα που ε, ζητούσε στην Αρκαζία στην Νότια Οσετία να υπάρξει ανάπτυξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά έγινε η επέμβαση εκεί. Για δεύτερη φορά να μην βρεθούμε πάλι μπροστά σε γεγονότα που δεν περιμέναμε. Έπειτα, ο κύριος Βανισβήλη, από ό,τι φαίνεται, θα ηγείται της χώρας από τα παρασκήνια. Είναι συνταγματικό να γίνεται αυτό χωρίς να έχει συνταγματικές ευθύνε. Έπειτα, Βανισβήλη ανοιχτά λέει ότι η αντιπολίτευση τώρα είναι κακή και θέλει να την αλλάξει από μια καλή, το Μουτζαρνάτσε. Το κόμμα Μουτζαρνάτσε προχωράει με τα μέσα ενημέρωσης, με αλλαγές από υπέρ της Ευρώπης σε λιγότερο υπέρ της Ευρώπης και η Γεωργία τελικά θα ακολουθήσει το δρόμο της Αρμενίας. Είναι ένα σενάριο αυτό πιθανό, έτσι το βλέπετε. Ευχαριστώ. Ο πρέσβης να απαντήσει δεν είναι βέβαια ακρόαση, έτσι, με τον πρέσβη της Γεωργίας, αλλά να απαντήσετε παρακαλώ κύριε πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Σάριος Βόλσκι για την ερώτησή σας. Εννοείται ότι δεν μπορώ να σας πω στα σίγουρα τι σκέφτονται οι διάφοροι παράγοντες στη Γεωργία. Το σενάριο το οποίο περιγράφεται δεν είναι απίθανο. Όμως ελπίζω ότι πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία τελικά θα αποφασιστεί βάσει των επιδόσεων των διαφόρων παικτών στην πολιτική σκηνή της Γεωργίας. Εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε βέβαια την απόφαση του εκλογικού σώματος, την σημειώνουμε απλώς. Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι είναι οι πιο υποστηρικτές της ευρωπαϊκής προσέγγισης στη Γεωργία θα ενισχύσουν την θέση τους. Κατόπιν τούτων. Ανταλαμβάνομαι ότι ελοχεύουν κινδύνοι και ακριβώς γι' αυτό τόνισα και νωρίτερα ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την δικιά μας δυνατότητα να επηρεάσουμε τα πράγματα, ώστε να καταστήσουμε ξεκάθαρο πως η επιτυχία της γεωργίας όσον αφορά την προσέγγιση προς την Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί. Με κάθε σεβασμό Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε με τον κατάλογο μιλητών. Ο κύριος Κόβαλ είναι ο πρώτος. Διαδικαστικό. Παρακαλώ κύριε Νέης. Ναι, ναι, έχω εδώ ένα διαδικαστικό. Μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η εξέλιξη. Πώς εργαζόμαστε δηλαδή σήμερα το απόγευμα. Φυσικά χαίρομαι και εγώ για την παρουσία εδώ του πρέσβη και τον ευχαριστώ, τον πρέσβη Δημητρόφ <clears throat> και όχι Κύριλοφ όπως κατά λάθο είπε αρχικά κυρία Νέης. Ναι, κάποιος συνάδελφος είναι Κύριλοφ και εγώ τον έκανα πρέσβη, είδατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συζητάμε για την Γεωργία και πολύ καλά κάνουμε. Αυτή όμως η ανταλλαγή όπου ακούμε τον πρέσβη και μετά τον κύριο Σάρους Βόλσκι και μετά ακούμε μόνο την απάντηση του πρέσβη και κανένας άλλος δεν είναι σε θέση να παρέμβει στο διάλογο αυτό, είναι περίεργο. Εγώ θέλω να παρέμβω. Αν συζητάμε τη Γεωργία, πολύ ωραία να τη συζητήσουμε. Την παρουσία του πρέσβη, ευχαρίστω, αλλά όχι με τον τρόπο που έγινε. Διαμαρτύρομαι γι' αυτό. Ναι. Ο και μετά θα απαντήσω. Εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα, εκπλήσω με τη διαδικασία. Η παρουσία του πρέσβη, με κάθε σεβασμό, δεν προβλεπόταν. Και φοβούμε ότι καταλήγουμε να έχουμε μια κρόση για τη Γεωργία που δεν είναι ο στόχος της σημερινής συζήτησης. Έχουμε πολλά ερωτηματικά λοιπόν επί της διαδικασίας, Πρόεδρε. Η παρουσία του πρέσβη ανακοινώθηκε στην αρχή και κανένας δεν ε, είχε αντίρρηση. Ανακοινώθηκε στην αρχή ότι ο πρέσβης θα αναφερθεί στην κατάσταση στη Γεωργία και εγώ επίσης είπα ότι δεν πρόκειται για κρόαση για τη Γεωργία και τώρα θα περάσουμε στην γενική συζήτηση. Συνεπώς, συνάδελφοι, η Γεωργία αποτελεί μέρος της συζήτησης, βεβαίως. Εκτός μικροφώνου, κυρία Κοπά, δεν ακούγεται. Ανακοινώθηκε στην αρχή και εσείς δεν φέρατε αντίρρηση στην αρχή. Δεν είπατε ότι είσαστε κατά της παρουσίας του πρέσβη εδώ, οπότε δεν βλέπω γιατί διαμαρτύρεστε, αλλά Ωραία. Συνεχίζουμε. Κύριε Μπρόκ. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο πιο χαλαρά να το δούμε. Έχουμε εδώ μια έκθεση μπροστά μας που και τη γεωργία συμπεριλαμβάνει. Αλλά όχι μόνο τη γεωργία. Και έχουμε <clears throat> σήμερα την ευκαιρία να παρίσταται ο πρέσβης και είχε προαναγγελθεί αυτό. Δεν υπήρξε κάποια ένσταση αντίρρηση και τώρα μπορούμε να δραχθούμε τη ευκαιρία να ακούσουμε αυτά τα στοιχεία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που σε σχέση με την ημερήσια διάταξη έγιναν και δεν χρειαζόταν να έχουμε ένα έξτρα ξεχωριστό σημείο για την ημερήσια διάταξη. Στο πλαίσιο τη έκθεση αυτή μπορούν να τεθούν αυτά τα ερωτήματα και προ τον πρέσβη και να απαντηθούν και να τα δούμε αυτά. Και μπορεί και να συνεχίσει με τι παρεμβάσει του και μπορεί να παραμείνει ο κύριος πρέσβης ε, και μπορεί και να παρίσταται και δεν τίθεται κανένα θέμα εδώ. Και κατά τα άλλα η συζήτηση για την έκθεση Σαριούς Βόρσκι Παντσέρι μπορεί να συνεχιστεί όπως προβλεπόταν. Δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα. Εκτός αν πιστέψει κανείς ότι με τυπικές τέτοια με τυπικούς, ε, ας το πω έτσι, τυπικά επιχειρήματα διαδικαστικά μπορεί κάτι τέτοιο να το αποτρέψει. Είμαι όμως ευγνώμων για το ότι ο πρέσβης ακολούθησε το αίτημά μας που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είχε διατυπωθεί να τοποθετηθεί επ' αυτόν. Και ε, για τη χώρα που αφορά αυτή η δραστηριότητα και οι παρατηρήσεις μου φαίνεται ότι είναι πολύ σκόπιμο να καλυφθεί με αυτή την αφορμή. Δεν πρέπει να υπάρχει εδώ κάποια αφορμή, να έχει υπάρξει κάποια αντίρρηση ή ένσταση. Δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα εγώ σε σχέση με αυτό. Συμβαίνει καμιά φορά να έχει κανείς διαφορετικές πολιτικές απόψεις και πρέπει να δεχθεί αυτές τις διαφορετικές τοποθετήσεις. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του κυρίου Δημητρόφ. Έχει πολύ μεγάλες επιδόσεις που ε, κατάφερε να δημιουργήσει για την μετάβαση και της ε, μεταβατικής περίοδου ε, για την ε, Ουκρινία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά με τη δική του δραστηριότητα και πρωτοβουλίες κατέσαν εφικτά. Για πρώτη φορά να υπάρξει μια ειρηνική, ας το πω έτσι, μετάθεση της εξουσίας και χωρίς τριβές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι μας. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ. Και τώρα νομίζω δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μείνουμε περισσότερο σε αυτό το ζήτημα, να περάσουμε σε άλλο. Άλλο διαδικαστικό, κυρία Νέτση, παρακαλώ personal fact, as they Ένα προσωπικό σχόλιο. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι κατά της παρουσίας του πρέσβη. Ουδόλος. Δεν μου αρέσει αυτό που οργάνωσε ο κύριος Σάριος Βόλσκι. Δεν διαμαρτύρομαι για την παρουσία του πρέσβη. Κανένας δεν μπορεί να ελέγξει το Σάριος Βόλσκι. Σε παρακαλώ, Αμέλη, κατάλαβε το. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην καθυστερούμε, αλλά ας περάσουμε στις παρεμβάσεις. Γιατί αν θέλεις μπορείς να μείνεις. Αν θέλει κάποιος να απευθύνει ένα ερώτημα προς τον πρέσβη, είναι εδώ για να μας ακούσει και να απαντήσει ας πάμε στη γενική συζήτηση για το θέμα που μας απασχολεί και που είναι στη μέση διάταξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ότι εκπονήθηκε αυτή η έκθεση. Θα έλεγα, αν όλα αυτά τα θέματα τα δει κανείς για τα οποία γίνεται λόγος, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ξεχνάμε όμως ένα σημαντικό στοιχείο μεταξύ αυτών. Ότι υπάρχει κάποια κόποση σε σχέση με την, ε, ε, τις εξελίξεις αυτές. Υπήρξε η υπόσχεση ότι θα υπήρχαν ε, διευκολύνσεις θεωρήσεων διαβατηρίων για την Ουκρανία. Τώρα απουσιάζει αυτό το στοιχείο. Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία αλλά και για τη Μολδαβία. Δεν κατέστη εφικτό. Είναι όμως ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Ακριβώς σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής στο Βίρνιος διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο αυτό το ζήτημα και είναι πολύ πιο αποφασιστική σημασία από ότι κάποιες εμπορικές πτυχέ εμπορική σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει υπευθυνό πνεύμα ότι σε σχέση με αυτές τις, ε, το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίων κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε τα θέματα των ε, ελέγχων στα σύνορα. Μπορούν όλα αυτά ηλεκτρονικά να γίνονται και να εξετάζονται, να ελέγχονται τα έγγραφα στα σύνορα ηλεκτρονικά. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει στα σύνορα σήμερα. Νομίζω ότι υπήρξε ένα σεμινάριο ε, όσον αφορά ε, ίδρυμα πολιτικής ε, ενημέρωσης για τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων. Είναι αποφασιστική σημασία στο θέμα των διευκολυσεων θεωρήσεων διαβατηρίων να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες. Για χώρες όπως την Ουκρανία και τη Μολδαβία η όλη αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναρτάται και εξαρτάται από αυτό το θέμα. Αν θα πετύχουμε τα υπεσχημένα πριν από τα ζητήματα εμπορίου ή εμπορική σημασία. Πρέπει αυτά τα ζητήματα να αποσαφινιστούν όσον αφορά διευκολύνσεις ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Και όσον αφορά το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας εδώ στην Ευρωβουλή αυτό <clears throat> και όσον αφορά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές παραβλέπουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Κοπά. Κύριε Κοπά, ευχαριστώ. Θέλω να μιλήσω εκ μέρου του ε, σκιώδους εισηγητή που δεν μπορεί να παραστεί. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ε, αμφισβητείται από πολλού και είναι προς το συμφέρον μας να ακούγονται θετικά σχόλια γι' αυτά. Ε, είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα της, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικά θα πρέπει να αποφασίσουμε αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρεί, ε, εκφράζει θετικά ή αρνητικά ε, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ανάλογα με το ποιο είναι στην εξουσία σε αυτές τις χώρες, ανάλογα με το ανεφίλη του ή εχθρή του. Ε, και το χρησιμοποιώ ως εργαλείο για το διακομματικό παιχνίδι. Αυτά εκ μέρους του συναδέλφου μου και τώρα εκ μέρους μου. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ε, ε, νέες εξελίξεις, ειδικά στο Νότο, θα πρέπει να αποκτήσει νέα ορμή, θα πρέπει να προωθήσει δράσεις για την σταθερότητα και τη δημοκρατία στην Νότια Μεσόγειο. Ε, η κοινωνία των πολιτών γίνεται αισθητή και στις χώρες της νότιας ε, γειτονίας και της ανατολικής γειτονίας. Ε, ζητούν κράτος δικαίου, σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ελευθερία του λόγου, ε, τη σκεφτική ελευθερία, ελευθερία του σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ. και αυτές είναι ουσιαστικά θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υποστηριχθούν. Πρέπει να επαναλάβουμε επίσης ότι ε, αυτές οι αξίες είναι πίσω από τις μεταρρυθμίσεις αυτές τις χώρες. Ε, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν πολιτική δέσμευση και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολιτικές σχέσεις και οικονομικός και πολιτικός διάλογος. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, για τον Νότο, είναι σημαντικό για την Ένωση να έχει ουσιαστικά ουσιαστικά κονδύλια για την προστασία των μεταναστών και ε, προσφύγων με ιδιαίτερη έμφαση στι γυναίκες και τα παιδιά. Οι περισσότερες ε, μεταρρυθμίσεις που έχουν υποβληθεί δείχνουν τη σημασία που δίνει το Κοινοβούλιο σε αυτήν την πολιτική. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο αυτό το ψήφισμα να εμπλουτιστεί με τις τροπολογίες που ενισχύουν ε, τις παραπάνω απόψεις. Ευχαριστώ κύριε Κοπά ο κ. Λανσπέργης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Διάβασα την, ε, το σχέδιο της έκθεσης. Και έχει περάσει βεβαίω ε, κάποιο χρόνο από τη στιγμή που συντάχθηκε η, έκθεση. Επομένω, κάποια από αυτά που αναφέρει είναι πλέον ε, ξεπερασμένα από τι εξελίξει. Αν συγκρίνεται αυτά που μας είπε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, της Βενετίας για την Ουκρανία και αυτά που λέει η έκθεση, κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν στην έκθεση. Υπάρχουν και κάποια σημεία που θα ήθελα να υπενθυμίσω για την ε, Αρμενία, Συρία, όχι διορθώνει ο Μίλτης, όχι Συρία, Γεωργία. Για την πρόοδο στην Αρμενία. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόοδος για να υπάρξει αυτή η συμφωνία ε, σύνδεσης. Ε, όλες οι προϋποθέσεις της συμφωνία αυτής της σύνδεση δεν έχουν ε, υλοποιηθεί. Ε, μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για επίλυση των ε, παγωμένων συγκρούσεων. Αυτά δεν έχουν γίνει. Ε, επομένως, ε, θα πρέπει να καταδικάσουμε τις πρόσφατες αποφάσεις της αρμενικής κυβέρνησης να στραφεί προς την Ρωσία και να στρέψει τα νότα της προ εμά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα γεγονότα. Για τη Γεωργία. χρειάζεται να δούμε με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα στην ε, γεωργία. Ε, προσοχή για να μην υπάρξει περαιτέρω, ε, α, προκλήσεις, ε, καταπάτηση εδαφών, πέρα από αυτά που έχουν καταπατηθεί ήδη, και προσάρτηση εδαφών. Για τη Συρία. Πρέπει να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να ζητήσουμε πιο συγκεκριμένα να σταματήσει η σύγκρουση της Συρίας. Ε, πρέπει να καταδικάσουμε την χρήση θανατηφόρων αερίων ε, επί του αμάχου πληθυσμού και να ζητήσουμε να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Επίσης, Υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε συνέχεια για τα όπλα, ανησυχούμε υποτίθεται για τα όπλα, θέλουμε να διώξουμε τα όπλα από τη Συρία, αλλά δεν μιλάμε καθόλου για του δολοφόνους. Δεν τονίζουμε καθόλου την ευθύνη ε, των δραστών. Όλων αυτών που παίρνουν αποφάσει όλων αυτών που χρησιμοποιούν τα όπλα. Δεν μιλάμε καθόλου για αυτό το πρόβλημα. Όλους, για, ό, για όλους αυτούς που εξεντονίζουν ε, τους πυράβλους με τα αέρια, επίσης δεν γίνεται λόγος. Ευχαριστώ κύριο Σόλτ. Mr. Scholz. Scholz ε, παρακαλώ. Schulz, έτσι, Scholz. Ε, πολύ καλά. Μαραμ Θεοχάρος. Κυρία Θεοχάρους παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω πιστεί... Would you please use your headphones? I'm speaking in Greek. Thank Δεν έχω πιστεί ότι η Αρμενία έχει επιλέξει από μόνη της αυτό το δρόμο και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε ένα πολύτιμο στρατηγικό σύμμαχο στον Κάφκασο, ειδικά αν συνεχίσουμε αυτό που έχει πει ο κύριος Λατσπέρχης, να καταδικάσουμε τις αποφάσεις των Αρμενίων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κλίμα μέσα στο οποίο ζει ο αρμενικός λαός, την απομόνωση... Okay. πρέπει, πρέπει να λάβουμε υπόψη το κλίμα, τον εκφοβισμό, τον φόβο, τον τρόμο μέσα στον οποίο ζει ο αρμενικός λαός, τις απειλές που δέχεται συνέχεια. Πρέπει να αποσυνδέσουμε το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την ε, συμφωνία σύνδεση και αυτή η επιλεκτική ευαισθησία όσον αφορά την κατοχή εδαφών θα πρέπει επιτέλους να μην αφήνεται ως double standards να διαφοροποιεί τις αποφάσεις μας. Όσον αφορά τον... Δεν έχω πιστεί προσωπικά γιατί μέχρι και πολύ πρόσφατα που είχα συναντήσει τους αξιωματούχους της Αρμενίας, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό κλπ. Ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση τους να στραφούν προς την ε, ήταν στραμμένη, είναι στραμμένη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα πριν πάρουμε κάποια απόφαση και η έκθεση δεν πρέπει ακριβώς να οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να βοηθήσουμε την Αρμενία να ξαναγυρίσει στην τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ε, Όσον αφορά το πρόβλημα του Καραμπάχ, ναι, σίγουρα πρέπει να λυθεί. Αλλά α εφαρμόσουμε επιτέλου στην περίπτωση του Καραμπάχ το, το, τον χάρτη των Ηνωμένων Ελευθερών και ειδικά το άρθρο 2 για την αυτοδιάθεση των λαών. Νομίζω ότι με αυτό το ζήτημα θα κλείσει οριστικά αυτή η σύγκρουση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι συνάδελφοι σίγουρα παρακολουθούν πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα τα σχετικά με την πολιτική γυτνίασης. Τα ζητήματα που τίθεται εδώ όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις γείτονες χώρες του Νότου είναι η έλλειψη σταθερότητας στην κατάσταση εκεί. Και σήμερα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί και έχουν συμπεριληφθεί στις τροπολογίες δεν ισχύουν πια ή εν πάση περιπτώσει είναι εν μέρη ενισχύει διότι έχει αλλάξει η κατάσταση εκεί. Για το Λίβανο. Υπάρχουν ε, κάποιες ανακρίβειες. Ε, ήρθα από το Λίβανο και είχα και εγώ προτείνει μια τροπολογία για το κλείσιμο των συνόρων όσον αφορά τους πρόσφυγες ε, Παλαιστίνους και Σύριους. Δεν είναι σωστό γιατί έκλεισε για λίγο, άνοιξε μετά. Πάντως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λίβανο σήμερα είναι πρώτα απ' όλα παντελής έλλειψη πόρων για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ακόμα και για τον ΟΗΕ και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική διακυβέρνηση και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε ε, λύσει ακόμα. Είπαμε στο Κοινοβούλιο ότι θα έπρεπε να μπει στη δουλειά, αλλά δυστυχώς κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να το αναλάβει. Οπότε, μήπως πρέπει να ενημερώσουμε την έκθεση, μήπως πρέπει να κάνουμε μια προφορική τροπολογία, μήπως πρέπει να περιμένουμε την ολομέλεια. Είμαστε δηλαδή σε ένα στάδιο όπου καλά δεν μπορούμε βέβαια να τα αλλάξουμε όλα. Η κατάσταση όμως αλλάζει από μέρα σε μέρα. Επίσης, κύριε Λαμπέργη, ναι, λέτε να καταδικάσουμε τους ενόχους, τα χημικά όπλα κλπ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας ότι υπήρξε συμφωνία για τα χημικά όπλα σήμερα και ίσως να συμπεριλάβουμε και άλλα στοιχεία από αυτά που λαμβάνουν χώρα στο, στη ε, Νέα Υόρκη σήμερα. Συνεπώς, μέχρι την Ολομέλεια να ξαναδούμε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε προφορικές τροπολογίες. Πάντως, ενημερώνω τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να χτενίσουμε κάποια σημεία ε, παρά το ξέρω το έργο που έγινε από τον εισηγητή, η κατάσταση είναι αυτή που αλλάζει και αλλάζει σημαντικά από μέρα σε μέρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στήρ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω το έργο και των δύο εισηγητών και να τονίσω δύο ζητήματα που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνοχή στις εκθέσεις που υποβάλλουμε και να λάβουμε υπόψη μας στις τροπολογίες, κάτι που οι συγκεκριτές είπαν ότι θα κάνουν. Ιδιαίτερα μάλιστα εν ώψη των πιο πρόσφατων γεγονότων. Μετά το πρώτο σχέδιο δηλαδή μέχρι την τελική εκδοχή. Υπό το φως μάλιστα των τελευταίων ψηφισμάτων που είχαμε στο Στρασβούργο για την κατάσταση στην Αίγυπτο αναφέρουμε επιθέσεις κατά των χριστιανών και το ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει κάποιο ρόλο εκεί. Εγώ πιστεύω ότι τέτοιες τροπολογίες έχουν θέση εδώ. Κάτι άλλο τώρα. Σε αυτού του είδους συζητήσεις θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο συστηματική συζήτηση για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα τις πολιτικές και στα ανατολικά μας και ανωτίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν είναι μια απλή συσσόρευση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στις διάφορες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι στη Γεωργία και την Αρμενία για παράδειγμα χάνει σε επιρροή. Από την άλλη η επιρροή της Μόσχας ενισχύεται. Η Μόσχα επίσης παρεμβαίνει στο θέμα της Συρίας. Συστηματικά δηλαδή έχουμε κάποια άποψη για όλα αυτά τα θέματα ώστε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην έκθεσή μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι η δικιά μου πολιτική ομάδα είναι επικριτική όσον αφορά τον προσανατολισμό της πολιτικής γυτνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχουμε πει και στην περίπτωση των ε, γεγονότων με την Αραβική Άνοιξη. Γιατί έχουμε, είχαμε μάλλον συμφωνίες με το καθεστώς του Μουμπάρεκ και όχι μόνο και αλλού που ποτέ δεν αμφισβητήσαμε γιατί αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι οικονομικές ανταλλαγές και όχι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που εμείς όμως θέλουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες, το ίδιο κανονικά πρέπει να θέλουμε και για τους υπόλοιπους. Συνεπώς η πολιτική αυτή προσπαθεί να είναι μια συμφωνία σύνδεσης σε οικονομικές βάσεις. Και περιμένουμε να προχωρήσουν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες για να υπάρξει ελεύθερο εμπόριο. Όμως οι ιδιωτικοποίηση, η απορρίθμιση κτλ. έχουν σαν αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Οι αξίες μας πάνε πίσω δηλαδή, όπου το χωρούν τα κεκτημένα επίσης. Τι θέλουμε τελικά, τι θέλουμε να εξάγουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν συμφωνούμε. Εμείς θέλουμε συμφωνίες σύνδεσης που να βασίζονται στην αμοιβαιότητα προκειμένου να υπάρξει ένας χώρος ευημαρίας βάσει κοινών αξιών μεταξύ μας και που να μην τις επιβάλλουμε. Εμείς λοιπόν δεν τον βλέπουμε τον προσανατολισμό αυτόν. Επιπλέον από τις σχέσεις που είχαμε με τον Μπεναλή και τον Μουμπάρεκ, τα δύο καθεστώτα που σας είπα πριν, υπάρχουν κόκκινες γραμμές που πρέπει να βάζουμε και είναι η Δυτική Σαχάρα και η Παλαιστίνη είναι δύο άλλες περιπτώσεις. Βάσει αυτής της ε, φιλοσοφίας λοιπόν, η Δυτική Σαχάρα πρέπει να ξέρουμε ότι βρίσκεται σε κατοχή από το Μαρόκο, όμως η πολιτική γυτνίασης μπαίνει πάνω από τα κριτήρια αυτά και έχουμε συμφωνίε σύνδεση με το Μαρόκο. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση τη Παλαιστίνη. Δεδομένου ότι υπάρχει συστηματική κατοχή, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Γιατί τελικά δεν ενδιαφερόμαστε φαίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σήμερα οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρονται για την οικονομία, την απορρίθμιση που να εγγυάται τη συσσόρευση του κεφαλαίου. Γι' αυτό και εμείς υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Επειδή υπάρχει και σχέση μας με την Τουρκία, που μιλάμε για την ένταξή της. Στα κριτήρια πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας την κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το ότι υπάρχουν εκεί στρατιώτες. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται παρά το ότι έχει καταδικάσει το θέμα αυτό η διεθνής κοινότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω κάποια σχόλια για την πολιτική γετνίαση με τις χώρες νοτίως της Ευρώπης. Άκουσα και τον κύριο Παντσέρη. Η ιδέα της έκθεσής του είναι τις task forces να τις επεκτείνουμε και σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία. Εγώ λοιπόν έχω υποβάλει μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση που λέω ότι που μιλάει για τις χώρες που βρίσκονται εκτός του συστήματος αυτού. Τώρα πιο συγκεκριμένα. Παράλληλα με τις συμφωνίες ελευθέρωσης εμπορίου υπάρχουν και τα θέματα υποδοχής μεταναστών. Εδώ θέλω να αναφερθώ στη Μοσογειακή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια αυτό το όργανο έχει γίνει πολύ σύγχρονο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει, και η κυρία Άστον το έχει πει για την Ορδανία, πρέπει να παίξει πιο σημαντικό ρόλο για συγκεκριμένες χώρες. για την Αίγυπτο όντως πρέπει να προσαρμόσουμε την διατύπωσή μας. Είχαμε ένα ψήφισμα που αναφερόταν σε μια διαδικασία συμφιλίωσης και εγώ επέβαλα τροπολογίες ακριβώς για τη γλώσσα, για τη διατύπωση. Θα ήθελα να είναι κάπως πιο θετική η γλώσσα που χρησιμοποιούμε τόσο για το Μαρόκο όσο και για την ε, Αλγερία. Γιατί νομίζω ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα θετικά στην περίπτωση των δύο αυτών χώρων. Για παράδειγμα ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε παρατηρητές για τις εκλογές εκεί και ότι ξεκίνησαν και διαπραγματεύσεις για σχέσεις με την Αλγερία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κύριο Στάνοκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σχόλιο για κάποιο που αναφέρθηκε από την συνάδελφο κυρία Ελένη Θεοχάρους για την Αρμενία. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρούσα εχθές όταν έγινε η συζήτηση και αρκετά εκτενή συζήτηση για την έκθεση Πορέμα. Δα ο Τόμας δεν μπορούσε να είναι παρόν, μίλησα εγώ για λογαριασμό του, που υποστηρίζει στεναρά τη θέση που εσύ πρότεινε, Ελένη και μπορώ να σου διασφαλίσω ότι δεν αποκόμισα την εντύπωση από τα όσα ακούστηκαν ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο ή αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Ευρωβουλής ε, θα έστρεφε τα νότα και θα διαφορούσε για την Αρμενία ενώ έλαβε δυστυχώς υπό σημαντική πίεση κάποια απόφαση η Αρμενία ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι την έλαβε χωρίς πίεση ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας ώστε να μείνει η πόρτα ανοιχτή προς την προσέγγιση της Αρμενίας προς την Ευρώπη για συμμετοχή και εμπλοκή στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοιο και ένα θέμα από τους πράσινους εχθές για την ε, απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων κτλ και σε σχέση με το Ναγκόρνο Καραμπάχ η ομάδα σου και η δική μου δεν θα υποστήριζε ένα τέτοιο αίτημα μέσα στο πλαίσιο της ε, χαλάρωσης των θεωρήσεων διαβατήριων. Τώρα σε σχέση με το τι ε, συνέβαινε στην Αρμενία ήμουν ο πρώτος εισηγητής για την ENP όταν ξεκίνησε η προσέγγιση αυτής της ιδέας ήμουν ο μόνος εισηγητής τότε πιστεύω στεναρά ότι θα μπορούσε μια τέτοια πρόταση να μπορέσει να ισχύσει για όλες τις χώρες. Έπρεπε όμως να υπάρξει μια πολύμορφη αντιμετώπιση. Είδαμε ότι δεν γινόταν να ακολουθηθεί μια ενιαία τέτοια προσέγγιση και έπρεπε να ληφθεί μια διαφοροποίηση υπόψεων. Η Μολδόβα και το Μαρόκο βρίσκονται σε μια διαφορετική κατάσταση ε, όπως και σε σχέση με αυτά τα θέματα και για την, ε, το Μαρόκο και την ε, Αλγερία οι διαφορές τους είναι μεγαλύτερες ε, σήμερα και σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη που είναι ένας παγωμένος αραβικός χειμώνας και όχι Άνοιξη πλέον σε σχέση με την προσέγγιση της δημοκρατίας όπως την χαιρόμαστε στην Ευρώπη και η Ρωσία αφυπνίστηκε σε σχέση με τα θέματα της Ανατολικής Γειτονίας σε σχέση με κάποια θέματα εθνικών συμφερόντων και παρακόλλησε τις εξελίξεις εξελίξεις. Ευελπιστώ παρόλα αυτά ότι η Ουκρανία θα έχει την δυνατότητα έναντι της μικρότερης γεωργίας να παραμείνει πιστή στην πορεία προσέγγισης ε, της Ευρώπης. Παρότι υπάρχουν ε, αντίξοοι, ε, αντίθετοι άνεμοι που φυσούν από πλευρά της Ρωσίας για να παρακολουθεί αυτή η προσέγγιση και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και για την έκθεση 2005 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Μεσόγειο και την ε, πρωτοβουλία που είχε αναλάβει τότε η Γαλλία για αυτήν την ευρωμεσογειακή προσέγγιση πάντα φυσικά φυσικά μπορούμε να προσεγγίζουμε την προσέγγιση να υπάρχει ένα μέτρο που να ισχύει για όλους. Αλλά πιστεύω εγώ ότι χρειάζεται μια πιο ευέλικτη, ελαστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποίησεις και διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Και τα είχα κάνει και δύο φορές, όχι μόνο για τον Νότο και την Ανατολή, αλλά και τώρα βλέπουμε ότι εξειδικεύεται η γειτονική σχέση αναχώρα, πιο εξειδικευμένα προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη κάποιες αρχές ε, με το ότι υπάρχουν ε, με κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των χωρών αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιομορφίες των επιμέρους χωρών. Είναι ένα είδος λεμποδρομίας, ένα είδος ανταγωνισμού σε σχέση με το πώς θα μπορέσει αυτή η σχέση να εξελιχθεί υπέρ της μίας ή άλλης χώρας. Και πρέπει να πούμε ότι παραμένει αυτή η προσέγγιση ως θετικό στοιχείο και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως εισηγητές να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με τη δεδομένη αυτή κατάσταση. Και παρόλα αυτά ως προσέγγιση είναι κάπως προβληματική θα έλεγα παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετίζω το έργο των δύο εισηγητών, του κυρίου Σάρκους ε, Βόλσκι και του κυρίου Παντζέρη. Συνεργάστηκαν για να υλοποιήσω μια αδύνατη αποστολή σχεδόν. Όταν διαβάζουμε την έκθεση διαπιστώνουμε ε, πόσο πραγματικά είναι αδύνατη αυτή η αποστολή. Mission impossible. Επομένως, ε, έχουμε βάλει διάφορα πράγματα παράτερα μεταξύ τους. Ένα, μια παράγραφο για τη Συρία, που πραγματικά δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω έτσι πώς έχουν τα πράγματα. Διαβάζω αυτά που λέει ο Σάριος Βόλσκι για τη Γεωργία επίσης, όπου λέει ότι πρόσφατα έγινε σοβαρή παναχώρηση των δημοκρατικών κανόνων. Πραγματικά διαρωτώ με ποια ήταν η δημοκρατική ποιότητα αυτών των κανόνων πριν αλλάξει η κυβερνητική πλειοψηφία. Ήταν καλύτερα. Ε, επίσης, η Αίγυπτος είναι μοναδική χώρα για την οποία ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει την αρχή της αιρεσιμότητας. Για καμία άλλη χώρα δεν ζητάμε το ίδιο πράγμα. Αισθάνομαι λοιπόν πολύ αμήχανα. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Καταλαβαίνω δεν μπορώ να φτιάξω μια έκθεση με 20 και 30 σελίδες. είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε αυτό που κάνουν δυστυχώς οι δύο συνεισηγητές. Δηλαδή, με μία φράση, ας πούμε, για τη Μολδαβία ξεπετάμε το θέμα. Η Βερονίκ Ντεκέζερ μίλησε για τις δυσκολίες που έχουμε. Γιατί αλλάζουν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα τα πράγματα που αυτά που γράφαμε πριν ε, λίγες εβδομάδες δεν ισχύουν πια σήμερα. Και αυτά που λέμε σήμερα σε δύο εβδομάδες θα έχουν αλλάξει πάλι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ενδεικτικό της αδυναμίας να ασκήσουμε συνεπή και μοναδική και ενιαία πολιτική γειτονίας. Μιλάμε για τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές χώρες. Μιλάω και για τα ανατολικά μας σύνορα και για τα νότια σύνορά μας, όπου η πλειάδα των χωρών ε, είναι εντυπωσιακή και η ανομοιομορφία τους μεγάλη. Επομένως, το θάρρος των δύο συνεισηγητών είναι σημαντικό. Διαρωτώ όμως, πρέπει να αποφασίσουμε εδώ στην ομάδα τι θα κάνουμε με αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρέντα. Πολύ σύντομα. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για τη δουλειά τους. Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες. Είμαι πεπισμένος ότι θα φτιάξουμε λογικούς συμβιβασμούς. Απλώς παίρνω το λόγο για να πω ότι έχω επιφύλαξη απέναντι σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο για την Αρμενία. Τα έλεγα και χθες αυτά. Θέλουν δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια μας απέναντι στη χειρονομία της ε, Ρωσίας. Προφανώς είναι απαράδεκτη. Προφανώς είναι απαράδεκτο και το γεγονός ότι η Αρμενία στράφηκε προς τη Ρωσία και έστρεψε τα νότα σε εμά. Θέλουμε να κλείσουμε εντελώ τα μάτια στη συμμετοχή της Αρμενίας σε αυτό το πρόγραμμα ε, και στη χειρονομία που έγινε απέναντι στη Ρωσία. Επίσης έχω δισταγμούς για αυτό που είπε η κυρία Νέιτς, ότι η ιδέα του η Βανισφίλη να κατασκευάσει τη δική του αντιπολίτευση, αυτό δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό. Αναφέρθηκε αυτή η δήλωση του Ιβανοσφίλη πριν από λίγο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. η χειρονομία αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί απερίφραστα ως απαράδεκτη. Ο κ. Παντζέρη. Μία διευκρίνηση θέλω να δώσω. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Εμείς κάναμε μια πολιτική επιλογή, την οποία ε, υπερασπίζομαι με νύχια και με δόντια. Δηλαδή, να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για την πολιτική ε, γειτονίας. Να αποφύγουμε αυτό που συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε διάφορες θέσεις. Να αντιπαραθέσουμε δηλαδή την πολιτική γειτονία προς Ανατολά και προς Νότο. Και να προσπαθήσουμε μέσα στα όρια του εφικτού να κάνουμε και μια αξιολόγηση και μια αξιολογική κρίση και να έχουμε και μια ευέλικτη πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις ε, καθημερινές εξελίξεις. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να βασιστούν στου οικονομικούς πόρους που έχουμε, σε προγράμματα που προτείνονται και σκοπό θα έχουν να υποστηρίξουν μια πολιτική οικονομικής και κοινωνική ανάπτυξης, μια πολιτική κινητικότητας, ε, κυκλική κύριε Μον, δηλαδή πρέπει να έχουμε μια πολιτική κινητικότητα, αλλά για την τακτική, ε, για την νόμιμη ε, μετανάστευση. Δηλαδή να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, αλλά να γυρνάνε πίσω στη χώρα του και να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τη χώρα του και στην οικονομία τη χώρα του. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω επίση γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε την δημοκρατική μετάβαση στον Νότο, αλλά φαντάζομαι και στην Ανατολή. Να υπάρξει κράτο δικαίου, να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, αυτά είναι βασικά στοιχεία είναι βασικά στοιχεία μιας πολιτικής γειτονίας που νομίζω ότι πρέπει να επιβεβαιωθούν και να επικαιροποιούνται συνέχεια. Το no for more πρέπει να το μετριάσουμε γιατί μερικές φορές ε, δημιουργούνται εκεί αντιφάσεις. Υπάρχει και το θέμα της τακτικής και μόνιμης επικαιροποίησης. Και επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συχνά δρούμε με τρόπο άκαμπτο και δεν είμαστε χρήσιμοι. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με πραγματικότητες που στην ανατολική πλευρά αλλά και στην, ε, στους νότιους γείτονες αλλάζουν από μέρα σε μέρα, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια κοινή αξιολόγηση και μετά να προβλέψουμε και μια σειρά από επικαιροποίησεις. Δεν θα επανέλθω στις ε, τροπολογίες, είναι πολλές, αλλά επανέλαβα ότι γράψαμε λίγα πράγματα λόγω του ότι έχουμε περιορισμένο χώρο. Σίγουρα οι τροπολογίες μπορεί να εμπλουτίσουν αυτά τα λίγα που γράψαμε και, θα, και για την Αλγύρια και για την Αίγυπτο αλλά και για άλλες χώρες θα δώσουν έτσι μια εικόνα πιο ε, ολοκληρωμένη. Βέβαια υπάρχουν και τροπολογίες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές. Έτσι. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από γεωγραφία και που πιστεύουν ότι οι χώρες της Νοτιού Αφρικής πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσοχή, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις τροπολογίες, έτσι. Ε, η δουλειά που κάνουμε θέλω να πιστεύω ότι είναι σοβαρή και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να συνεισφέρει ε, στη διαμόρφωση μιας πολιτικής ε, γειτονίας ε, που να ευθυγραμμίζεται και να λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις στις χώρες αυτές, ανατολικά και νότια. Να βοηθήσει λοιπόν το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες λοιπόν θα τελειοποιήσουμε ακόμα περισσότερο μαζί με τον συνάδελφο Βόλφ και αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πρώτα ότι αυτό που είναι σημαντικό σε, αυτή τη δίδυμη, σε αυτές τις δίδυμες εκθέσεις είναι το γενικότερο μήνυμα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους να μην απολέσουμε το δάσος ενώπιον μας εστιαζόμενοι σε κάποιο δέντρο και είμαι βαθιά πεισμένος και κάνω λόγο και εξ ονόματος του συναδέλφου ότι υπάρχει <clears throat> μια ενδύναμη, ας το πω έτσι, ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιομορφίες ε, των κάποιων χωρών έναντι κοινών στοιχείων. Αλλά αν φανταστούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση και έχουμε μόνο ξεχωριστά περιπτώσεις όπως το Μαρόκο, την Αρμενία, την Αλγερία, πόσο πιο αποδυναμωμένοι θα είμαστε. Υπάρχει συνέργεια σε σχέση με την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί και μετά να εξειδικεύσουμε ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τις ανάγκες ατομικά των επιμέρους χωρών. Χρειάζεται λοιπόν ένα στεναρό, ας το πω έτσι, αμφίδρομα ικανό να δράσει ε, από πλευράς του ένα τέτοιο εγχείρημα ή σχέδιο ώστε να έχει η Ένωση ένα περίγυρο, ένα κλίμα ειρήνης, ε, ευημερίας, ασφάλειας ε, γύρω της, γύρω από τα σύνορά της. Αυτό είναι η κυριότερη πολιτική προτεραιότητα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, αυτή η έκθεση εσκεμένα δεν είναι εξειδικευμένη αναχώρα και αναειδιομορφίες χωρών. Αν θέλει κανείς τέτοιου είδους ε, συστατικά και χαρακτηριστικά ξεχωριστά, ας ανατρέξει στις εκθέσεις για τις επιμέρους χώρες. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί. Αυτοπεριοριστήκαμε και είμαι υπερήφανος ότι για τη Μολδόβα κατάφερα σε μια πρόταση να τα πω όλα όσα μπορούσα να πω. Όσο είναι, όσο είναι πιο σύντομο ένα κείμενο, τόσο είναι και πιο αποτελεσματικό. Και γιατί κανείς δεν έχει χρόνο να διαβάζει εκτενή κείμενα. Έτσι λοιπόν, οποίο θέλει λεπτομέρειες αστραφής στις εκθέσεις που αφορούν εξειδικευμένα τις επιμέρους χώρες σε λεπτομέρειες. Για κάποια θέματα που δεν είναι δυνατόν να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους, σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και θα το κάνω αυτό. Αλλά για τον κύριο Λαντσμπέργης. Κύριε Λαντσμπέργης, θα υπάρξουν προφανώς μεταβολές σίγουρα και όσον αφορά και την Αρμενία και την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η κατάσταση μετεξελίσσεται ούτως ή άλλως. Για την κυρία Νέιτς δεν βρίσκεται, δεν παρευρίσκεται η κυρία Νέιτς πλέον, έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Και το γεγονό ότι διακόπτει ο μιλήτης. Εντάξει, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι πιστεύω ότι αλλάζει ο σημερινός πραγματικός κόσμος και αυτός, αυτό δεν είναι λόγος να μην προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα πράγματα ή να τα προσεγγίσουμε. Οι τελικές διατυπώσεις ε, θα πρέπει να γίνουν στο τέλος μιας τέτοιας μετεξέλιξης και αν δεν γίνει κάτι δεν πάει στραβά στο νότο τότε και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να είμαστε όσο το δυνατόν πιο επίκαιροι θα υπάρξει επικαιροποίηση για τις ε, μεταβολές αυτή είναι η απάντησή μου προς τον κύριο Λαντσμπέργης προς την κυρία Νέιτς τώρα επικαιροποίηση λοιπόν και με την επικαιροποίηση αναφέρθηκα ήδη σε αυτήν για τη γεωργία αυτό... Διαπιστώνω αυτό που λέτε για την υποχώρηση της δημοκρατίας στη Γεωργία. Υπάρχει έκθεση Αλεσμπέρκ. Για μένα είναι λεπτό το θέμα, αλλά περιγράφει την υποχώρηση των προδιαγραφών της δημοκρατίας στην ε, έκθεση αυτή. Τώρα για τον κύριο Κόβαλ. Είναι εδώ είπε πόσο σημαντικό είναι το θέμα των θεωρήσεων. Και εδώ όμως, σας είπα, λέμε στην έκθεση ότι θα πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση θεωρήσεων και η προοπτική για ένα σύστημα χωρίς θεωρήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι μια οριζόντια και συνοπτική έκθεση. Λοιπόν και πάλι σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε. Να ξέρετε ότι οι παρατηρήσεις σας είτε γραπτές είτε προφορικές θα περάσουν από επεξεργασία. Θα τις σκεφτούμε, θα τις επεξεργαστούμε σίγουρα και ο κύριος Παντζέρη και εγώ. Και προσβλέπουμε στην στήριξή σας. Ιδιαίτερα γι' αυτό το γενικό μήνυμα που είναι μια δοκιμή για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί αν αποτύχει αυτή η πολιτική μας για την γυτνίαση, φανταστείτε τι θα γίνει με την γενικότερη πολιτική μας. Τι Είναι μια πολιτική η οποία φτιάχτηκε κάπως βιαστικά, οπότε δεν θα συμφωνούσατε με αυτό το κάπως ε, προκλητική σκέψη που ακούσαμε ότι η όλη αυτή η πολιτική έγινε υπό την πίεση κάποιων χωρών μελών που δεν θέλανε να ενοχλήσουν την Ρωσία, που θέλανε να προσφέρουν μια εναλλακτική ε, προπτική ένταξη της Ουκρανίας. για να γίνει δηλαδή μια ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία. Πάντως ιστορικά κοιτώντα τα πράγματα, πράγματι νομίζω ότι έτσι τα βιαστικά φτιάχτηκε αυτή η πολιτική για να κρατήσει τις χώρες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε παρά το όσα λένε ο κύριος Σέρους Βόλσκι και ο κύριος Παντζέρη, Νομίζω ότι πρόκειται για μια αντίδραση στην γεωπολιτική κατάσταση που επικρατούσε πριν από 8-9 χρόνια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εξακολουθεί να ισχύει δεδομένων των γεγονότων. Είναι πολύ αμφίβολο αν εξακολουθεί να ισχύει η κατάσταση που είχαμε και τότε. Να δούμε, οι ιστορικές μνήμες είναι σωστές. Αυτό το είδους ιστορική μνήμη πάει πριν και από αυτά το, οποίο αναφέρεται ο κύριος Τάνοκ. Κι εγώ τότε ήμουνα σε αυτή την κατάσταση. Οπότε πρέπει να δούμε τα πράγματα από δύο διαφορετικές προοπτικές. Δεν είναι μόνο ιστορική προοπτική. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλώς έγινε. Θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα, αλλά καλώς έγινε. Αν δεν είχε γίνει θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Λέτε στα βιαστικά. Ε, καλύτερα αργά παρά ποτέ, θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, θα ήταν καλύτερα, αλλά βλέπετε η πολιτική είναι η τέχνη του να κάνεις το maximum κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν ονειρεύεστε μια πολιτική γειτονία η οποία θα αντικατασταθεί από την πολιτική διεύρυνση, ακόμα και αν συμφωνώ μαζί σα, θα απαντήσω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό σήμερα. Οπότε καλύτερα μια πολιτική γειτονία παρά τίποτα. Πολλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Και όταν λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και διαδραστική κλπ. κλπ όλα αυτά, αυτό ακριβώς δείχνουν. Υπάρχει μια ολόκληρη παράγραφος εδώ η οποία λέει ότι συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα έπρεπε να είναι α, β, γ, δ κτλ. Πολλά θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, να διορθώσουμε, αλλά να θέτουμε υπό αμφισβήτηση την ίδια αυτή την πολιτική χωρίς την οποία η εξωτερική πολιτική της Ένωσης θα ήταν περίπου ανύπαρκτη, ε, είναι υπερβολή. Αν είναι γιατί έχετε περισσότερε φιλοδοξίες, εγώ είμαι μαζί σας. Αλλά προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με αυτό που έχουμε, αντί να το αμφισβητούμε από τη ρίζα του, γιατί είναι μια ουσιαστική πολιτική που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. λίγες παρατηρήσεις η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ε, επινοήθηκε από του Πολωνούς και Σουηδούς ε, φίλου μα ώστε θεσμικά οι σχέσει με αυτέ τι χώρε να ενισχυθούν σε, σαν μια, α το πω έτσι, πρώιμη φάση στην ε, ευρωπαϊκή του ένταξη. Και έτσι πρέπει να ανοίξουν δρόμοι για να μπορέσει να πορεθεί η Ουκρανία προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το ιστορικά σημαντικό σε, αυτή την, σε αυτό το εγχείρημα. Δεύτερο, βλέπω το πρόβλημα το οποίο έχουν οι συνάδελφοι, οι αυτή η έκθεση δηλαδή που είναι γενικά μια γενικότερη έκθεση να, ότι βρίσκεται μέσα σε μια φάση μεταβολών και διαρκών αλλαγών. Είναι μια έκτακτη ξεχωριστή κατάσταση. Το να βρούμε μια συνετή λογική οδό που θα πορευτούμε είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να έχουμε την έκθεση ως ε, είχε προσεγγιστεί. Τώρα, αν στο τέλος ε, θα προσυπογραφεί και θα εγγραφεί, ε, θα μονογραφηθεί η συμφωνία αυτή σε σχέση με την Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία κτλ. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει σε σχέση να κριθεί από τις συγχρονίες, τις χρονικές εξελίξεις ώστε να υπάρξει ένα ελαστικό πλαίσιο για να επιτευχθεί ώστε να μην ληφθούν αποφάσεις που θα είναι πρόημες και πρόορες πριν από την ώρα τους βιαστικές, να αναμείνουμε να οριμάσουν τα πράγματα ή ε, να έχουμε και την έκθεση Κβασνιεύσκη για παράδειγμα που θα αναμείνουμε να ε, κατατεθεί. Δεν έχω ακόμα διαμορφώσει τελεσίδικα την άποψή μου. Ξέρω αυτό που επιθυμώ, να προσυπογράψω και να εγκρίνω. Δεν, δεν ξέρω ακόμα αν θα το καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί ή όχι. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτά τα θέματα. Το βρίσκω καλό τις ηγητές το θέμα με την νότια γειτονία αλλάζει και αυτό καθημερινά στις συνιστώσεις του. Δεν έχουμε εμείς να λάβουμε αυτή την απόφαση ναι ή όχι, υπέρ ή κατά, σε σχέση με σύνοδο κορυφής του Βίνιους. Πρέπει να ξαναδούμε τι τις ανάγκες ε, που είναι ξεχωριστές ε, σε σχέση με αυτό. Παρακαλώ να συνεχιστεί, να αφήσουμε να συνεχιστεί η διαδικασία, αλλά με ανοιχτό πνεύμα και πλαίσιο. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι για παράδειγμα στο τέλος πριν από την λήψη απόφαση στην Ολομέλεια θα μπορούσαμε να συνέρθουμε ώστε να δούμε αυτή τη μία πρόταση, μία διατύπωση από την οποία θα εξαρτηθούν τα πράγματα να, να την εξετάσουμε. Ίσως όμως μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι αναγκαίο αυτό και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για παράδειγμα σε σχέση με την Ουκρανία. Πολλά πράγματα εξελίσσονται λογικά και συνετά ώστε μπορεί να δει κανείς το φως ε, ε, να προσεγγίζει στην άκρη του τούνελ ώστε να εγκριθεί. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε το benchmarking σε σχέση με τα θέματα δικαιοσύνης να διασφαλιστεί με ένα λογικό τρόπο. Δηλαδή τα θέματα για παράδειγμα της έκθεσης Κβασνιεύσκη να μπορέσουν λογικά να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν διότι το θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης είναι πολύ σοβαρό και απομένει και η περίπτωση Τιμοσέγκο Τώρα να δούμε αν αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί και πώς. Και σε σχέση με την παρέμβαση στην Γιάλτα για παράδειγμα τέθηκε ένα κέριο ερώτημα και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Και ελπίζω και σήμερα το πρωί το ανέφερα σε σχέση με τις συζητήσεις ε, που γίνονται και με την Προεδρία, τη Λιθουανική Προεδρία, ότι βλέπω δηλαδή με άλλα λόγια ότι υπάρχει η πολιτική βούληση. Είναι εφικτό με την πολιτική βούληση και με τον προβληματισμό αυτό να προχωρήσουμε και από πλευρά ε, του Πρόεδρου Γιαννουκόβιτς ε, σε σχέση με μια δημόσια συνάντηση με την ε, Πρόεδρο Ριουμπασκάιτε είπε ότι δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αυτό το θέμα, δεν έχει ληφθεί τελεσίδικη απόφαση. Αυτό το βρήκα αξιοπρόσεκτο σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του και πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την τάση ή πορεία ώστε εδώ οι πλειοψηφικές θέσεις που θα δημιουργηθούν στο Κοινοβούλιο και που είχαμε στο Κοινοβούλιο να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να αποσαφινιστούν ώστε και πέρα από αυτό το πλαίσιο να μπορέσουν να αξιολογηθούν αυτά τα πράγματα και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει. Και ελπίζω ότι η ρωσική στάση τις επόμενες εβδομάδες και μήνες όσον αφορά την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Ήταν αντιπαραγωγική η στάση της Ρωσίας. Το συζητήσαμε σήμερα το πρωί το θέμα με την έκθεση ο Σάλιβαν. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προθυμία, για παράδειγμα, για το θέμα προθυμίας υπογραφής της συμφωνίας με την Ουκρανία. Φυσικά αυτό αφορά και τη Οδαβία και τη Γεωργία και άλλες απαιτήσει Μολδαβία και Γεωργία. Ως Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τις χώρες εκείνες που πρέπει να τύχουν υποστήριξη ώστε να αντέξουν, αντέξουν στην πίεση που ασκείται από αυτές. Πρέπει να υπάρχει αυτή η προθυμία όσον αφορά τις διεργασίες και το όφελος και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ώστε να υπάρξουν χρηματοοικονομικές δυνατότητες που θα επιτευθούν και θα χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει ιδιαίτερα έντονα τους επόμενους, ε, τις επόμενες εβδομάδες να εξετάσουμε τα θέματα τα ενεργειακά και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ενεργειακά θέματα προς αυτές τις χώρες. <clears throat> και όπως έχουμε την έκθεση που υπάρχει σχετικά η βούληση για την διασύνδεση για τα ενεργειακά θέματα έχει τεράστια σημασία ώστε αυτές οι χώρες να αντιμετωπίσουν ένα ψυχρό χειμώνα και να μπορέσουν να ε, νιώσουν και να ζήσουν, να βιώσουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που θα τις συνδράμει και θα τις υποστηρίξει. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα αναγκαία ώστε να μπορέσει ο στόχος να επιτευχθεί. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο εισηγητές. Τι είπατε εσείς? Äh, ναι και τον κύριο Δημητρό φυσικά σας ευχαριστούμε θερμά ότι είχατε την υπομονή να προσέλθετε και μας δώσατε τις ε, αναγκαίες χρήσιμες πληροφορίες ε, από πλευρά σας και σε σχέση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας κάποια πράγματα δεν έχουν επιτύχει το επίπεδο εκείνο το οποίο θα επιθυμούσαμε και υπάρχουν και ανησυχίες θα επισημάνατε κύριε Πρέσβη είναι θεμητά τα, θεμητές οι ανησυχίες μας αν παραμείνουν όμως τα πράγματα ως έχουν και συνεχιστούν έτσι θα μπορούμε ίσως ε, να δούμε τη δυνατότητα μονογραφής αυτής της ε, συμφωνίας, ώστε η μονογραφή αυτή να μπορέσει να υποστηριχθεί και μετά οι διαδικασίες μεταρρύθμισης στη Γεωργία να μπορέσουν, ε, όπως και σε σχέση με την Ουκρανία τα έχουμε συζητήσει, να πετύχουν την επόμενη φάση, το επόμενο βήμα, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στη φάση υπογραφής της συμφωνίας με την Γεωργία. Εδώ και από πλευρά συνδρομή τη Επιτροπή είναι σημαντική υποστήριξη. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν. Και περνάμε τώρα στη δική μου έκθεση για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Θα είμαι πολύ σύντομος αν συμφωνείτε. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να συζητηθούν. 340 τροπολογίες έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας, για τις τροπολογίες σας, για τις νέες ιδέες για τις οποίες θα προβληματιστώ επ' αυτών <clears throat> και ένα μεγάλο αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών έχω έχουμε ε, εκπονήσει που ότι αύριο ή μεθαύριο θα μπορέσουμε να σας τις διαθέσουμε. Να σας τις διαθέσουμε όπως έλεγα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τις δικές σας παρατηρήσεις και τοποθετήσεις στην έκθεση. Θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας ότι δηλαδή τα κύρια μηνύματα κλειδιά αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε και Κάποιες από τις ιδιομορφίες ε, ε, για τις επιμέρους χώρες και για τις επιμέρους περιοχές ή περιφέρειες ε, να μπορέσουμε να καταλήξουμε έτσι σε κάποια γενικά συμπεράσματα. Μην απαριθμίσουμε ξεχωριστά κάθε χώρα μεμονωμένα. Παρότι μπορεί να είναι η μέθοδος αυτή ίσως πιο σωστή, πιστεύω πρέπει να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία που πρότεινα στην αξιολόγηση των χωρών αυτών γιατί κάθε ένας φυσικά έχει μια χώρα που πρέπει, θέλει επ' αυτής να εστιαστούν όλοι. Αλλά διαφορετικά κανείς δεν θα μπορέσει να διαβάσει την έκθεση αν έχει τόσο μεγάλη έκταση και θα πάει χαμένο το μήνυμα και ο κόπος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε έτσι να πορεθούμε να οδεύσουμε σε μια οδό που θα ε, συμφωνήσετε κι εσείς επ' αυτής. Έχουμε την διεύρυνση της εταιρικής σχέσης Ρωσία και άλλα που έχουμε συμπεριλάβει στην πρώτη φάση του κειμένου και πρέπει να προσπαθήσουμε κατά την επόμενη εβδομάδα να βρούμε μια χρονική στιγμή με τους σκιώδεις εισηγητές να συζητήσουμε για αυτές τις, ε, τις ε, συμβαστικές τροπολογίες κατά την αρχή της επόμενης εβδομάδας ώστε να έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες προς ψήφιση και έγκριση ώστε στις 9 Οκτωβρίου χωρίς κόπο και χωρίς ε, προβλήματα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε προς έγκριση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα και σε σχέση με τις τροπολογίες αυτές θεωρώ <clears throat> ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε αν είμαστε αποτελεσματικοί να πετύχουμε αυτό το στόχο. Εντάξει. Ωραία, 9 Οκτωβρίου λοιπόν. Ο Σίλβιο ομολόγησε ότι είναι, έκανε, έγινε ένα σφάλμα. Καινούριο και αυτό από πλευρά του. Η 7η Οκτωβρίου είναι, όχι η 9η Οκτωβρίου. Εντάξει, 7 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε προσέγγιση. Κυρία Κοπά, παρακαλώ ο κύριος Πάσκος και ο εισηγητής μας μιλάει σε μια διεθνή διάσκεψη και εγώ μπορώ να παρουσιάσω διάφορα σημεία για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην έκθεση εκ μέρους του. Όπως είπαμε στην αρχική μας συζήτηση, εκτιμούμε την στρατηγική προοπτική της έκθεσης, Υποστηρίζουμε, θα υποστηρίξουμε τις ε, Τρει χειρόγραφες τροπολογίες και θέλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο συνεκτικέ. Οι τροπολογίες θα πρέπει να συμπληρώνουν το κείμενο γενικά και να μην προσθέτουν περιττές τροπολογίε. Η ομάδα μου θα ήθελε να προωθήσει μια ισορροπημένη θέση για τα πιο πιεστικά θέματα της ε, ΚΕΠΑ. Ε, ε, προσβλέπουμε στην, ε, στις συμβαστικές τροπολογίες του κ. Μπροκ. Οι τροπολογίες του S&D ε, των σοσιαλιστών επαναλαμβάνουν κάποια πολιτικά θέματα σημαντικά. Η ε, ενίσχυση της διατλαντικής ε, εταιρικής σχέψης με την προστασία της νομοθεσίας και την προστασία των δεδομένων. Μια σφεκτική προσέγγιση, η υποστήριξη ουσιαστικών αποφάσεων στην σύνοδο του Δεκεμβρίου για την άμυνα, δράσεις, πιέσεις στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, και σημασία της αρχής ε, της ευθύνης. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά με τον ε, εισηγητή για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε στη διάθεσή σας εμείς οι φιλελεύθεροι για να συζητήσουμε τους συμβιβασμούς. Θα ήθελα να κάνω τρία σημαντικά σχόλια. Πρώτον, απέχουμε λίγες βδομάδες από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να εντείνουμε την πίεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το Συμβούλιο δηλαδή, για να επωφεληθούν από αυτή την ανευπροηγουμένου ε, ευκαιρία που έχουν να συζητήσουν ε, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Άκουσα σχόλια της ε, διαφόρων πρωθυπουργών που είπαν ότι δεν περιμένουν και πολλά να προκύψουν από αυτή τη συνδοκορυφή. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο. Να προσπαθήσουν επίση να φτάσουν σε μία συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που σημαίνει την επίλυση του Κυπριακού, Δεύτερον, να βρούμε ένα τρόπο για να αναθεώρηση της ΚΠΑ. είχαμε όλα τα κρατημέλη ζήτησαν μια ε, ζήτησαν, είπαν μάλλον ότι να βρούμε ε, παραπέρα από αυτό που πρέπει ε, το να έχουμε μία λευκή βίβλο. Εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η γειτονιά μας, και το συζητήσαμε πολύ προηγουμένως, καταλαβαίνει το πώς εννοούμε εμείς τον πλουραλισμό και τα πρότυπά μας και τους κανόνες μας. όχι μόνο για τη δημοκρατική εκλογή των εκπροσώπων μας, αλλά και το πώς γίνεται δημοκρατική διακυβέρνηση. Σεβασμό της αντιπολίτευσης και με σεβασμό της διαφωνίας. Αυτά τα τρία ουσιαστικά θέματα θα ήθελε η ομάδα μου να συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Και από δική μου πλευράς και πλευράς των Πρασίνων φυσικά, ευχαρίσω στην επόμενη εβδομάδα να συνέρθουμε μαζί σας, να δούμε τις συμβαστικές τροπολογίες, να δούμε ποιες θα, τι μπορεί να γίνει. Κάποια σημεία θα ήθελα να αναφέρω που από δική μας πλευράς ε, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά και παρακαλούμε να τα συμπεριλάβετε. Για το ένα συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Νταφ, τη σπουδαιότητα δηλαδή της διεύρυνσης, της επέκτασης. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα και εργαλεία που έχουμε για να μπορέσουμε υπό το πρίσμα της ειρηνευτικής, ε, ειρηνικής και ειρηνευτικής πολιτικής να σημειώσουμε πρόοδο. Θέλω να σας ζητήσω να δεχθείτε μία από τις τροπολογίες μας όπου με κριτικό πνεύμα αντιμετωπίζουμε την δυνατό, τις δυνατότητες για τα Δυτικά Βαλκάνια, για κάποιες χώρες για παράδειγμα όπως τη Μακεδονία, τι μπορεί να γίνει, διότι αν δεν γίνουν αυτά παρακολύεται η πολιτική μας σε αυτή την περίπτωση και τις σχέσεις, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τις ΗΠΑ Είναι πολύ αναγκαίο πιστεύω εδώ να το θέσουμε αυτό το θέμα για την κριτική που ασκείται για τις ε, περιπτώσεις ε, ε, κατασκοπίας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. Δοκιμάζονται ιδιαίτερα σκληρά οι σχέσεις της ΕΕ με τη ΣΥΠΑ και αυτό πρέπει να ενταχθεί στην έκθεσή σας ως θέμα πιστεύω. Και ένα ακόμα θέμα, το Ιράν. Θα έλεγα ότι ακριβώς με τα πιο πρόσφατα στοιχεία και τις πιο πρόσφατες κινήσεις του νέου Προέδρου του Ιράν έχει νόημα να αναφερθούμε στο θέμα του Ιράν. Και εκεί έχουμε μια πρόταση, μια τροπολογία και ελπίζουμε ότι ευμενώς θα την αντιμετωπίσετε και θα την συμπεριλάβετε θα την υπαγάγετε στην έκθεσή σας. Και ένα ακόμα στοιχείο. Λόγω των επίκαιρων γεγονότων πρέπει να επισημάνουμε ότι από ευρωπαϊκής πλευράς θέλουμε να αποφύγουμε ευρωπαϊκές εταιρείες να κάνουν dual use, δηλαδή να έχουν μηχανισμούς ε, σύλληψης, για παράδειγμα μηχανισμούς ε, χρήσεις ε, που μπορούν να τύχουν διτής χρήσης από αυταρχικά καθεστώτα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ευρωπαϊκές εταιρείες να παράγουν τέτοια προϊόντα και να τα διαθέτουν σε αυταρχικά καταστατικά καθεστώτα. Είναι κάποια από τα σημεία που είναι πολύ σημαντικά για μας. Θα έπρεπε νομίζω με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθείτε και να εγκρίνετε αυτά τα θέματα να ενταχθούν στην έκθεσή σας ώστε να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να καλυφθούν. Ευχαριστώ. gospodine Evo samo vrlo kratko s obzirom da su i drugi kolege spomenuli. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. είμαι πολύ σύντομο γιατί οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα Δυτικά Βαλκάνια και στη διεύρυνση. Δεν θα πω περισσότερα από αυτά που είπαν εκείνοι, αλλά να σας θυμίσω μόνο ότι είναι ακριβώς αυτές τις περιοχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται, υπάρχουν αποτελέσματα. Σερβία, κοσυφοπεδιο Οπότε αυτό που θέλω να σας πω επ' αυτού είναι ποιες είναι οι προσδοκίες για το μέλλον. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πολιτική απέναντι στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Ο Επίτροπος Φίλε συναντάει όλους τους πολιτικούς ηγέτες ε, όπου να είναι από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στις 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα θα υπάρξει μια πολιτική συζήτηση εδώ στην Επιτροπή αυτή θα έπρεπε επίση να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει επίσης ότι προχωράει. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, αν δεν μπορούμε να πετύχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, ε, ας ξεχάσουμε τότε την Ευρώπη ως παγκόσμιο παίκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για αυτό το θέμα θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι κάπως ασυνήθιστο για τέτοιες εκθέσεις ε, για την εξωτερική πολιτική και εξωτερική πολιτική ασφάλειας. Ε, όμως ήρθε η χρονική στιγμή θα έλεγα όπου θα ήταν σωστό και νόμιμο να πούμε το εξής. Η υγεία η υγεία πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη και αυτή να καλύπτεται ως στοιχείο που αφορά την ασφάλεια. Και μάλιστα ανάλογα με τα όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο παγκόσμια. Η Υγεία λοιπόν. Και σε σχέση με αυτό το θέμα του πώς δηλαδή ποια είναι η κατάσταση υγείας των ανθρώπων και πώς έχει επιδεινωθεί για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι θα έλεγα ένα θέμα στρατηγικής σημασίας και σπουδαιότητας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν θα ήταν δυνατόν η δική μου τροπολογία να ληφθεί υπόψη από εσά, Πρόεδρε. Με ακούτε, να ληφθεί υπόψη από εσά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς συζητάμε αυτή την εποχή μια έκθεση η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή για τις τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει. Η έκθεση αφορά όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές υποθέσεις. Έχει να κάνει επίσης και με θέματα τα οποία συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ. Θέματα τα οποία επίσης ε, προσέχουν πάρα πολύ οι πολίτες μας. Αυτή η διάσταση της νότιας εταιρικής σχέσης πρέπει να ευθυγραμμιστεί και με άλλες εκθέσεις, ώστε να στείλουμε ένα και μοναδικό μήνυμα προς τις εν λόγω χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί και ένα ακόμα θέμα στην έκθεση και είναι το εξή. Το θέμα της, επο... της ε, παρακολούθησης από το των Ηνωμένων Μιλάμε επίσης για τις θεωρήσεις και για τις τροποποίησεις που πρέπει να γίνουν στο θέμα αυτό των θεωρήσεων. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις ήταν επικοδομητικές. Θα ξαναδώ αυτές τις τροπολογίες. Σε ποιο βαθμό μπορούν συνολικά να ενταχθούν στην έκθεσή μου, ώστε ας το πω έτσι να διασφαλιστεί η ισορροπία των συστατικών στοιχείων της έκθεσής μου. Και γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος κ. Νταφ όσον αφορά τη λευκή βίβλο, το λευκό βιβλίο. Ένα λευκό βιβλίο είναι φυσικά μια αντανάκλαση των θέσεων των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ευαισθησιών τους. Πρέπει όμως να είναι ταυτόχρονα και μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Γι' αυτό δεν επαρκεί μόνο με ε, κρατικές ε, θέσεις των κρατών μελών ε, να συντίθεται από αυτήν. Πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία που θα απορρέει και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι Άλλο θέμα είναι το θέμα του Λευκού Βιβλίου. Πρέπει να βρούμε λοιπόν διατυπώσεις, τέτοιου είδους διατυπώσεις που να διευκολύνουν για παράδειγμα το πώς η βρετανική επιφύλαξη και προφύλαξη σε τέτοια θέματα θα μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αντανακλάται. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια συνετή λογική θέση. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Είπα ότι αύριο ή μεθαύριο θα μπορέσουν να αποσταλούν οι τροπολογίες, οι προτάσεις. Είμαστε πρόθυμοι αν και πριν από συνάντησή μας τη Δευτέρα ή Τρίτη, έχετε κάποιες παρατηρήσεις, αν ξέχασα κάτι κτλ, να έχουμε διμερώς άμεση επαφή, ώστε να μπορέσουν κάποιες ε, προτάσεις να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε απήχηση και να εγκριθούν. Ευχαριστώ θερμά. Αν ναι, μπορείς να αναλάβεις εσύ την ε, Προεδρία για μια στιγμή, για ένα μικρό διάστημα. Uh, uh, Συνεχίζουμε συνάδελφοι και περνάμε στην γνωμοδότηση όσον αφορά τις ε, εγγύησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την κάλυψη ζημιών δηλαδή από χρηματοδοτικές δραστηριότητε που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης. Η συγητής μας, μάλλον συντάκτης γνωμοδότησης, είναι ο συνάδελφος Γιάτσεκ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 Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εξωτερική μας πολιτική και προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Στόχος μας λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εποπτεύουμε την βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ω συζητητή, λοιπόν έχω διαπιστώσει τα εξή που θέλω να βάλω στην έκθεση. Είναι πρώτον να συνάδουν όλα με το άρθρο 21 της Συνθήκης Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βασικό η ΕΤΕ να διασφαλίζει ότι κάθε οικονομική τη δραστηριότητα συνεισφέρει και συμπληρώνει την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποσαφηνίζει. Οι δραστηριότητέ τη πρέπει να συνάδουν με τι αρχέ δηλαδή εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ευχαριστώ του σκιώδει συζητητέ και του ευρωβουλευτέ ε, τους υπόλοιπους οι οποίοι ενισχύουν την ε, γνωμοδότησή μου τις απόψεις τους. Δεύτερον, έχω συμπεριλάβει τροπολογίες οι οποίες υπογραμμίζουν ε, περισσότερο σε βάθος συνεργασία με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, προκειμένου να υπάρξει ε, συμπληρωματικότητα. Έπειτα, διαφάνεια. Το έχουν πει και άλλοι εισηγητές. Υπογραμμίζω επίση τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης λέω ότι η ΕΤΕ πρέπει να ε, συζητάει με όλους τους ενδιαφερόμενους και οι αποφάσεις της να διέπονται από διαφάνεια. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή Προπολογισμών συζήτησε ήδη στις 18 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά όταν ο κύριος Καλφίν, ο εισηγητής, πρότεινε να αυξηθεί το ανώτατο όριο κατά ένα δις ευρώ για να φτάσει η εντολή στα επίπεδα των 30 δισεκατομμυρίων συνολικά. Ενώ τώρα είναι 25 για σταθερά και υπάρχουν και άλλα τρία για την περίοδο μέχρι το 2013. Πιστεύω ότι πρέπει να δεχτούμε την πρόταση αυτή. Κυρίως γιατί πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες που είναι προς ένταξη και ο δανεισμός έχει αυξηθεί πολύ από την αρχή της εντολής. Συνεπώς, Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω από τους εκπροσώπους της ΕΤΕ να μας πούνε ποιες είναι οι προοπτικές της ε, τράπεζας αυτή τη στιγμή και τι γίνεται με τις ανάγκες επενδύσεων στις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά μας, αλλά και νοτίως, δεδομένης μάλιστα και της κρίσης στην Αίγυπτο και τη Συρία. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει τη δυνατότητα να αυξήσει την αρρωγή της με τις στόχους και με την ποσά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες και τους ευρωβουλευτές για τη συνεισφορά τους, για τις τροπολογίες τους, ιδιαίτερα από την Άλτε, του κ. Βότσον, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, από την κυρία Γιακονσάρη και από τους Πρασίνους του κ. Μπουτικόφερ που στηρίζουν βασικά και συμπληρώνουν τη γνωμοδότηση αυτή. Κάποιες όμως από αυτές πρέπει να τις συζητήσουμε παρετέρω. Θα προσπαθήσω να καταλήξω σε συμβαστικές τροπολογίες και θα λάβω όλα, υπόψη μου όλα τα σχόλιά σας τα σημερινά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ΕΤΕ, λοιπόν, να μας πει τι μπορούμε να απαντήσουμε στον εισηγητή μας, στον συντάκτη της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Προτασέβιτς για αυτή τη γνωμοδότηση από πλευράς του και για την συνεργασία που είχαμε σχετικά, διότι θεωρούμε ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση. Στρέφομαι αμέσως στην ουσία του θέματος. Πιστεύουμε ότι ο κυριότερος στόχος των δραστηριοτήτων μας είναι ουσιαστικά να υποστηρίξουμε τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ένα επαρκές επίπεδο επενδύσεων όσον αφορά το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο μπορούμε να δίνουμε πιστώσεις, δάνεια και θα φτάσουμε στο όριο του σχεδόν 30 δις ε, όσον αφορά όλες τις περιφέρειες ε, συνολικά. Αυτό το επίπεδο μπορεί να διασφαλιστεί και στο επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με τις επενδύσεις στον δημόσιο τομέα και για τις δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές ιδιαίτερα όσον αφορά και την προένταξη ή και την ε, πολιτική γειτονίας. Ε, σε σχέση με την πρόταση αυτή θα συνεπαγόταν ιδιαίτερη επίπτωση σε σχέση με την γειτονία μας, ενώ η δράση μας μπορεί να υποστηρίξει και την σύγκληση όσον αφορά ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ευρωπαϊκές πολιτικές που ε, σε σχέση με τις χώρες αυτές που θέλουμε να προσεγγίσουν προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σε σχέση με μια ενιαία προσέγγιση. Στη νότια γειτονία ζητήθηκε να υποστηρίξουμε τη μεταβατική περίοδο αυτών των χωρών που προοδεύουν προ οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσει και μπορούμε με επαρκή βιώσιμα επίπεδα να το διασφαλίσουμε στην ανατολική γειτονία. Σταδιακά αυξάνουμε τι δραστηριότητε μα στο χρονικό αυτό διάστημα από το 2007 θα επιτύχουμε φέτος πάνω από ένα δις 1,2 δις επενδύσεων στις, ε, στις χώρες αυτές. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με αυτή την τάση, ώστε να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές και μελλοντικά. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στους διάφορους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτος που θα λάβει τον λόγο είναι η κυρία Λίσα Γιακονσάρη, παρακαλώ, από τους σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία Γιακονσάρη, σας ευχαριστώ πολύ Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης ε, και το σχέδιο έκθεσης έχουν θετικές βάσεις, θετικά θεμέλια και είναι ισορροπημένες οι προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε <clears throat> σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή κονδυλίων να δούμε ποιες προσαρμογές μπορούν να γίνουν αν αφαιρέσουμε από κάποια χώρα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμιση. Αν αυξηθεί για κάποια χώρα αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα κονδύλια από κάποια άλλη χώρα. Κάποιος παίρνει παραπάνω και πάντα αυτό γίνεται εις βάρος, όταν παίρνει κάποιος περισσότερα κονδύλια, εις βάρος κάποιου άλλου. Όμως, εν πάση περιπτώσει, μια αύξηση σε σχέση με την ανατολική γειτονία για την εντολή αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε με ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη οροφή 25 δις συν επιπλέον 3 δις ώστε στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί. Συμφωνώ με την έκθεση ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε κάποια θέματα. Πρώτον, τα δικαιώματα του ανθρώπου, θεμελιώδεις ελευθερίες, δημοκρατικές αξίες και αρχές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και διατάξεις που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαβρωθούν, δεν θα υπονομευθούν όλα αυτά μέσω άλλων δράσεων. Γι' αυτό οι χώρες που θα σέβονται και θα προσαρμόζονται με αυτές τις αρχές θα πρέπει να λαμβάνονται ξεχωριστά υπόψη και για τις χρηματοοικονομικές δράσεις ε, που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές ε, που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υποστηρίζουμε έτσι την εφαρμογή αυτών των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων και διεθνών <clears throat> συμφωνιών ακόμα και των συμφωνιών και συμβάσεων για τις ε, περιβαλλοντικές αλλαγές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα άλλο σημαντικό θέμα όπως ε, ακούστηκε μόλις είναι και η διαφάνεια και η δημοσιοποίηση στοιχείων προς ε, τους πολίτες και πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε με την πρόσφατα εγκριθήσα ε, έκθεσή μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες προδιαγραφές για να αντιμετωπίσουμε και να προφυλαχθούμε εναντί της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ομάδα τώρα <clears throat> της Άλντε Watson και μετά εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγχαίρω το Γιάτσεκ για την έκθεσή του. Ε, νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουμε και αυτό φαίνεται από τις τροπολογίες που υποβάλαμε. Μιλάμε για 25 δις, πολλά λεφτά. Για 7 χρόνια, έτσι. 25 δις για 7 χρόνια. Εάν επιτύχει όμως ο κ. Χόιερ ε, και μέσω της επιστολής που έγραψε τον κύριο Μπρόκ μπορεί το ποσό να, να ανέβει σε 30 δις για 7 χρόνια. Πολλά λεφτά. Και οι τροπολογίες που ε, προσπαθούν να αυξήσουν τη διαφάνεια σε αυτές τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία, να βοηθήσουμε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στον κόσμο και προσπαθούν επίσης τον εξωτερικό δανεισμό της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων να την ευθυγραμμίσουμε με τους στόχους που έχουμε εμείς καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, προσθετού περιβάλλοντος κτλ. Ερώτηση τώρα. Θέλουμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόσφαση στα έγγραφα να εφαρμοστεί πλήρως. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην είναι ε, διαφανής ε, και να έχει τη δική της πολιτική διαφάνειας. Θέλω να ρωτήσω την τράπεζα γιατί δεν είναι έτοιμη, όπως προτείνει μία από τις τροπολογίες μου να δημοσιεύσει πλήρως τις συμφωνίες τις οποίες ε, έχει με τρίτες χώρες. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η δημόσια πληροφορία, η πληροφορία αυτή προς το κοινό, σε ό,τι αφορά την ισορροπία. Γιατί τόσο πολλά λεφτά πάνε στη Λατινική Αμερική και τόσα λίγα στην Ασία. Γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, μεγαλύτερη αναλογικότητα ανάλογα και με τον πληθυσμό που έχουν αυτές τις περιοχές. Ε, υπέβαλα λοιπόν σχετικές τροπολογίες για να αλλάξει η... ο λόγος αυτός, το κλάσμα αυτό. Επίσης, γιατί η Ταϊβάν αντιμετωπίζεται σαν χώρα ε, απέναντι όπως την Κούβα, ε, το Αφγανιστάν και η Λευκορωσία που έχουν κυρώσεις, δηλαδή και όχι όπως το Κοσφοπέδιο και η Σιγκαπούρη και γιατί τη βάζουμε στον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών, γιατί θεωρούμε ότι είναι χώρα υποκυρώσει. Σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση με άλλε ευρωπαϊκές πολιτικές, οι προτάσει μου στι τροπολογίε 42, 62 κτλ. είναι ο δανεισμό να γίνεται με βάση τις αρχές της ευρωπαϊκής Νομοθεσία. Η απάντηση τη τράπεζα είναι ότι αυτό δεν είναι εφικτό ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν ισχύει ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δέχομαι αυτό. Εγώ δεν λέω να γίνει με βάση την νομοθεσία, αλλά με βάση τις αρχές της νομοθεσίας. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να ζητάω κάτι τέτοιο. Και δεν θα πρέπει να πετάμε λεφτά για, σε προβληματικά καθεστώτα για την ε, κλιματική αλλαγή. Ε, 22-23% των ποσών του ποσού του εξωτερικού ε, δανεισμού ε, πηγαίνει για προγράμματα καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Εγώ λέω να φτάσει στο 40%. Ε, η τράπεζα μου λέει δεν γίνεται. Τι είναι το εφικτό ποσοστό, 30-35%. Επίσης, προγράμματα για το φυσικό αέριο. γιατί τα, υποστηρίζουμε. Οι εταιρείε φυσικού αερίου βγάζουν δισεκατομμύρια δολάρια ε, σε κέρδη. Ε, μπορούν να χρηματοδοτήσουν τους δικούς τους αγωγούς. Γιατί εμείς να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά για, το κλιμα... για την κλιματική αλλαγή. Για... Να... Γιατί να μην ε, χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά για να περάσουμε σε πράσινες ενέργειες. Και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, τις οποίες δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, αλλά θα ήθελα λιγάκι η τράπεζα να μας απαντήσει με σοβαρό τρόπο σε, αυτά τα προ... σε αυτούς τους προβληματισμούς που έχουμε. Και εν πάση περιπτώσει αυτή η έκθεση πρέπει κάποια από αυτά τα θέματα να τα θέσει. Ευχαριστώ. Η Σαμπίνη θα κάνει την επόμενη παρέμβαση. Μετά θα απαντήσει η τράπεζα και ο πρόσωπο της Κομισιόν. Είναι μια γνωμοδότηση για μια έκθεση για την ευρωπαϊκή εγγύηση για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικέ δραστηριότητε. Επομένως, το πεδίο της έκθεσης είναι πολύ πιο στενό από αυτό το πολύ ευρύ επί του οποίου εσεί ε, τοποθετηθήκατε και σχολιάσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Εξ ονόματο ε, της αριστερής ε, <clears throat> κομματικής ομάδας έχω κάποιε τροπολογίε και θα ήθελα σύντομα να πω περθύνως πρόκειται και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αφενός πιστεύουμε ότι περαιτέρω είναι απαραίτητο προγράμματα για την πολιτική ανάπτυξη να υποστηριχθούν. Μια και όχι μόνο ιδιωτικά αλλά και κρατικά δημόσια τέτοια προγράμματα και σχέδια πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Γενικά όπου πρόκειται για τις δημόσιες ή κρατικές υποδομές που αφορούν τα θέματα υγείας και τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Να υποστηρίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε οι στόχοι της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών να μπορέσουν να επιτευχθούν, όπως αναφέρεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και μια αντίστοιχη τροπολογία που έχουμε καταθέσει. Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Ένα από τα θέματα πυρήνες, ε, κύρια θέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση και να υποστηριχθεί τροπολογία μας όσον αφορά την ε, ε, έγκριση κονδυλίων ή ε, κατανομή κονδυλίων δεν θα πρέπει αποκλειστικά να υπάρχει η δυνατότητα μόνο σε αυτό το όργανο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα λάβει τον λόγο τώρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Παρακαλώ να είναι το σύντομο, όσο δυνατόν πιο σύντομος. <clears throat> Το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχουμε τον αρμόδιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου ανάμεσά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Λαμπρινίδη τα θέματα της αρμοδιότητάς του μαζί του. Και πρέπει να προετοιμάσουμε και την αίθουσα και για το γεγονός ότι θα έχουμε και μια και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση που θα διεξαχθεί. Δηλαδή πιέζει πραγματικά ο χρόνος ασφικτικά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρώτη, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ τους κοιόδη συζητητές για τις τροπολογίες τους. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός. Και μπορούμε να δούμε και τα θέματα επιμέρους και χωριστά, αν θέλετε. Για την πρόσβαση στα έγγραφα εφαρμόζουμε την σύμβαση IRUS, και σε όλες τις δραστηριότητες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το λέω να αμφισβήτητα. Έχουμε την πολιτική διαφάνεια όμως γιατί πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μας ως τράπεζα. Παράλληλα όμως ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουμε όλες τις πολιτικές πρόσβασεις στα έγγραφα. Για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, είναι συμφωνίε πλαίσιο που δημιουργούμε, που συνάπτουμε με χώρες εταίρους, που καλύπτουν την διπλωματική ασυλία και την, το πλαίσιο δραστηριοτήτων μας στις τρίτες χώρες αυτές. Δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερα πολιτικό αυτές οι συμφωνίες. Δεν έχουμε πρόβλημα επίσης να σας τις δώσουμε αυτές τις συμφωνίες. Απλώς υπάρχουν πολλές που έχουν υπογραφεί όλα αυτά τα χρόνια και χρειαζόμαστε και την συμφωνία του άλλου μέρους για να δημοσιεύσουμε αυτές τις συμφωνίες. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από μόνοι μας. Ε, και το άλλο μέρος, το συμβαλλόμενο μέρος, πρέπει να συμφωνήσει για τη δημοσιοποίηση ε, των συμφωνιών. Τώρα, γιατί τόσα λεφτά, πολύ περισσότερα λεφτά στην ε, Λατινική Αμερική και λιγότερα στην Ασία. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι ανάγκες όλων των περιοχών του πλανήτη είναι τόσο ψηλές ε, για την ανάπτυξη του ε, ιδιωτικού τομέα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανανεώσιμες ενέργειες, ε, δημόσιο τομέα, υγεία και εκπαίδευση ενδεχομένω. Σε τόσε πολλέ χώρε στον κόσμο έχουμε τόσε ανάγκε. Α, και κλιματική δράση βέβαια. Που μακάρι να είχαμε και τα δεκαπλάσια από, αυτά, από τα ποσά που έχουμε για κάθε περιοχή. Το βασικό είναι να ακολουθήσουμε τις ε, πολιτικές προτεραιότητες, ε, όπως διαμορφώνονται από τα ευρωπαϊκά όργανα. Εμείς δεν έχουμε καμία προτίμηση. Ανάλογα με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εμείς κινούμεθα. Το ίδιο για την Ταϊβάν. Είναι πολιτική απόφαση αυτή. Εμείς δεν κάνουμε την επιλογή να τη βάλουμε στον α ή το β κατάλογο. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ας αποφασίσουν ποιες χώρες είναι επιλέξιμες και ποιες δεν είναι. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, φυσικά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε καμία από τις νομοθεσίες μας πέραν των συνόρων μας για τις προμήθειες, για το περιβάλλον, για τα πρότυπά μας. Απλώς προσπαθούμε να προωθήσουμε τα δικά μας πρότυπα για το περιβάλλον, για τις προμήθειες, για την ε, μη συμμόρφωση κάποιων ε, χωρών. Φυσικά αυτό πρέπει να γίνει με ανάλυση αναπρόγραμμα. Και με βάση την εμπειρία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθούμε απλώς να προωθήσουμε ε, τις αξίες μας ε, στους, στις επενδύσεις μας στο εξωτερικό. Απλώς δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε αυτές τις αξίες. Δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε όπως επιβάλλουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το περιβάλλον τώρα. Το 25% είναι ένα στόχος που έχει καθοριστεί από το Συμβούλιο μας για όλες τις επιχειρήσεις της τράπεζας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, λογικό είναι να έχουμε το ίδιο ποσοστό ε, και για τις επιχειρήσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το 90% των δραστηριοτήτων μας είναι στην, Ευρωπαϊκή Ένωση και το 10% εκτός. Με βάση την εντολή που έχουμε, έχουμε, έχει προβλεφθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Είμαστε άνετοι με αυτό το ποσοστό. Το να το ξεπεράσουμε θα, πρέπει, θα, θα σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τις επιλογές μας στους άλλους στόχους. Για τα προγράμματα φυσικού αερίου. Αυτό είναι θέμα επιλεξιμότητας. Όσοι λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις, αποφασίσουν και για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Και τώρα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λίγα σύντομα σχόλια. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή σας. Τα σχόλιά σας μας είναι πολύ χρήσιμα, τα σημειώσαμε όλα. Θέλω όμως να επανέλθω σε ένα ζήτημα που νομίζω ότι έθεσε ο εισηγητής για το συνολικό προπολογισμό, το συνολικό ποσό και τι σημαίνει αυτό οικονομικά. Τα 52 δισεκατομμύρια ανώτατο όριο έχει τεθεί από ένα ταμείο εγγύσεων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Οπότε προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι 9% της συνολικής εντολής καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύσεων. Αν λοιπόν το μέγεθος αυξηθεί και πάει από τα 25 στα 30 δισεκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν και περισσότερα κονδύλια μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο Αυτοεγγύσεων. Δεν έχω το ακριβές ποσό, θα προσπαθήσουμε πάντως να κάνουμε τους υπολογισμούς έγκαιρα πριν γίνει συζήτηση την Πέμπτη στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σύντομος. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ανταλλαγή αυτή απόψεων για το σημαντικό αυτό θέμα σας ευχαριστούν επίσης. Υπενθυμίζω ότι 10 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Τώρα, έληξε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στην ε, συνομιλία που θα έχουμε με τον κύριο Λεμπρινίδη. Πρόκειται όμως για μια συνάντηση που γίνεται και κλεισμένο το θυρών. Γι' αυτό παρακαλώ όποιος δεν δικαιούται να βρίσκεται στην αίθουσα, παρακαλώ να αποχωρήσει. Πρέπει και εγώ να λείψω για λίγα λεπτά.